Bene. Καλώς ορίσατε. Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Επίτροπο Ναυράτσης που είναι εδώ σήμερα μαζί μας και τους τέσσερις ε, πρέσβεις ε, για την ευρωπαϊκή αφήγηση, του οποίου θα σας συστήσω και φυσικά και τα μέλη που είναι παρόντα. Θα συνεχίσω στα Ιταλικά. Έχουμε το προνόμιο να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα μας, επομένως επειδή έχουμε και εξαιρετικούς διερμηνείς, μπορούν να σας βοηθήσουν. Φορέστε τα ακουστικά σας. Έτσι θα είμαι και πιο λακωνική και πιο σαφής. Ωραία λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Φορέστε όλοι ακουστικά. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την ε, συνάντηση την οποία επιθυμούσαμε διακαώς και μάλιστα γίνεται και σε μια σημαντική ημέρα. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής σήμερα, επομένως θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό να συζητούμε και μια ευρωπαϊκή αφήγηση που έχει και μια μουσική νότα, διότι η Ευρώπη χωρίς τη μουσική είναι μια ιστορία χωρίς ε, το κατάλληλο soundtrack, ε, την κατάλληλη ηχητική υπόκρουση. Επομένως ε, θα συζητήσουμε για αυτή την αφήγηση με μια μουσική νότα. Έχουμε εδώ και τον συνάδελφο, ο οποίος ε, ήταν και στην ε, Επιτροπή Πολιτισμού πριν από κάποια χρόνια, ο συνάδελφος Λόκεκαρτ. Δεν σας βλέπω, Άννα, εκεί είστε. Και ήταν αυτός ο οποίος ε, προωθούσε την Επιτροπή Πολιτισμού. Ε, τώρα βέβαια έχει αναλάβει άλλη αποστολή για να ξεκινήσει το 2003, αυτό το, 13, συγγνώμη, αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα για την Ευρώπη και τον πολιτισμό. Το 2015 είχαμε κάποιες προπαρασκευαστικές δράσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν και το 2016 και σύν το χρόνο μετατράπηκε σε μια πολιτική που δεν είναι τόσο μια πολιτική για τον πολιτισμό στην Ευρώπη, αλλά ε, ένα ε, τρόπος να δώσουμε μια πολιτιστική προοπτική στην Ευρώπη δεν θεωρούμε τόσο πολύ ότι πρέπει να έχουμε πολιτικές, αλλά αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε η Ευρώπη σήμερα είναι να έχει μια προοπτική ταυτότητας, πολυφωνίας, κοινών αξιών και να είναι ανοιχτή προς τον υπόλοιπο κόσμο. Αν θέλουμε να είμαστε παγκόσμιοι παράγοντες ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ε, έχουμε και ε, πολιτιστικό έργο και να βοηθούμε και τις ανταλλαγές ε, με τις νέες γενναίες και να τους κληροδοτούμε ε, ως μαρτυρία τον πολιτισμό μας ε, ως Ευρώπη που φαίνεται σήμερα να χάνει την ταυτότητά της, το ρόλο της, ακόμα και την αλληλεγγύη της δυστυχώς. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα πραγματικότητα και μια νέα αφήγηση. Αυτό το σχέδιο λοιπόν ε, έχει και συμβολικό χαρακτήρα και θέλουμε να έχουμε κοινού ε, ψυχήτε και σώματε την Ευρώπη για να μπορέσουμε ε, να έχουμε διάφορους τομείς, έχουμε τον πολιτιστικό, τον επιστημονικό τομέα, τον τομέα της δημιουργίας που έχουν συγκεντρωθεί για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πριν από τις εκλογές του 2014 ε, παρουσιάστηκε αυτή η δήλωση και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι εκεί υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ε, φράση ότι η Ευρώπη είναι μια ψυχική κατάσταση κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα και μια τεράστια ευθύνη. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική φράση, διότι μας αποδίδει ευθύνε για το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο πολιτισμός, αλλά και το ρόλο που πρέπει να έχει ο ίδιος ο πολιτισμός ε, εντός των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αποφασίσαμε λοιπόν να ε, παρακολουθήσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, να έχει μια συνέχεια το παραπαρασκευαστικό πρόγραμμα και σε αυτή την πρώτη φάση ο Επίτροπος ε, Ναυράτσης θέλησε να ανοίξει και τις πόρτες ε, για μια πιο γενική και πιο ευρεία συζήτηση στην οποία θα συμμετέχουν ιδιαίτερα και οι νέες γενιές και αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό με δημόσιες συζητήσεις και στα κράτη-μέλη αλλά και στα μέσα κοινωνικής ε, δικτύωσης. Ε, υπήρχε και συμμετοχή κάποιων βουλευτών για να μπορέσουμε να δούμε ε, πώς θα μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο και τι θα πρέπει να γίνει στη συνέχεια. Να υπενθυμίσω ότι ξεκίνησε αυτό το στάδιο το Φεβρουάριο του 2016, δηλαδή πριν από μερικούς μήνες, παρουσία φοιτητών του Erasmus νέων, ασκουμένων και υπάρχει αυτή η νέα φιλοσοφία που θα μας υποδείξετε εσείς ε, και αφορά και μια κοινότητα, αν θέλετε, αυτών των νέων ανθρώπων που μπορούν να είναι και πρωταγωνιστές ε, στη συζήτηση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ε, να μην είναι μόνο θεατές ε, το κοινό στο οποίο αποφθηνόμαστε, αλλά να είναι και οι πρωταγωνιστές της Ευρώπης. Ε, συμφωνώ απόλυτα με αυτό το σκεπτικό και πρέπει επίσης να αντιληφθούμε ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα μας διευκρινίσετε εσείς καλύτερα, το οποίο απευθύνεται σε διάφορους τομείς και πρωτίστως θα έχουμε και τις μεγάλες προσωπικότητες, τις διανόησεις, ε, καλλιτέχνες, και ερμηνευτέ τη ευρωπαϊκή δημιουργικότητα, του ευρωπαϊκού πολιτισμού και τη μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά που έχει η Ευρώπη, αλλά θα αποτελήσουν και προγεφύρωμα με του νέου, ε, κάτι το οποίο έλειπε στο πρώτο στάδιο. Εγώ δεν θα πω περισσότερα, γιατί εσεί θα πρέπει να μα τα πείτε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ. Και έχουμε και τους τέσσερις ε, πρέσβεις. Έπρεπε να είναι έξι, αλλά οι δύο είχαν κάποιο πρόβλημα και δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Ε, μετά λοιπόν από την παρέμβαση του Επιτρόπου θα τους δώσουμε το λόγο. Είναι η Πάτρικ Κόβαξ που είναι ο πρόεδρος ε, της ε, Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Νέων Επιχειρηματών, ο Μάικολ Κλάιμπερ, ερευνητές, πρώην μέλος της Ακαδημίας Επιστεωμών της Πολωνίας. Σνέσκα, γιατί το επίθετό σας είναι πολύ περίπλοκο. Σας ξέρουν όλοι ο ε, Σνεύσκα, Σνεύσκα Μιχαήλοβιτς, είναι εκπρόσωπος του η δική μας Ευρώπη και ο Πολ Τζαρντάν, πασίγνωστος, που είναι ο πολύ δραστήριος Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Μποζάρ ε, των Βρυξελών. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα λοιπόν. Δεν συμβαίνει συχνά να έχουμε ένα πάνελ τέτοιου επίπεδου και τόσο με διαφορετικής εκπροσώπησης. Έχουμε πάντα ε, πολλούς συνομιλητές στην Επιτροπή μας, αλλά τώρα έχουμε πρωταγωνιστές του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Λοιπόν, θα κάνουμε ε, αυτά που σας είπα. Έχουμε περίπου μια ώρα για να συνεισυζητήσουμε. Για 10 λεπτά να δώσω το λόγο λοιπόν στον Επίτροπο Ναυράτσιτς για να μας ε, ε, περιγράψει το νέο στάδιο αυτής της στρατηγικής, αυτής της νέας αφήγησης και ε, θα δούμε και ένα βίντεο. Στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στους τέσσερις πρέσβεις και από εκεί και πέρα θα ακούσουμε και τους συναδελφούς ε, εάν θέλουν να λάβουν το λόγο. Έχετε το λόγο, Επίτροπε Ναυράτζιτς. Ευχαριστώ, <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ και ευχαριστώ την Σίλβια Κώστα που μας δίνει την ευκαιρία να προβούμε σε άμεσο διάλογο μαζί σας για το νέο αφήγημα, το νέο ευρωπαϊκό αφήγημα. Είναι και σωστός ο τόπος για να μπούμε σε αυτή τη δεύτερη φάση του νέου αφηγήματος, του νέου ευρωπαϊκού αφήγηματος, διότι η πρωτοβουλία αυτή έχει τις ε, ρίζεστε στην Επιτροπή σας, στο έργο της Επιτροπής σας. Το 2013 ζητήσατε να δημιουργηθεί ένα έργο, ένα project, το οποίο θα φέρει την Ευρώπη κοντά στους πολίτες της, τονίζοντας τις κοινέ πολιτιστικές αξίες που μας καθορίζουν ως Ευρωπαίους πολίτες πέρα από τα σύνορα. Η αρχική αυτή πρωτοβουλία που έλαβε την μορφή ενός πιλωτικού προγράμματος και την οποία ακολούθησαν πολλές συζητήσεις με συμμετοχή εξεχουσών προσωπικότητων όπως τον Ντόναλτ Τούσκ, τότε Πρωθυπουργό της Πολωνίας, τον Ερή Κολέτα, Πρωθυπουργό της ε, Ιταλικής Δημοκρατίας, τη Γερμανίδα Καγκελάριο και τον πρώην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χουέν Μανουέλ Μπαρόσο. Αυτά τα πρόσωπα είχαν συμμετάσχει στις συζητήσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν σε μια διακήρυξη που αποκλήθηκε το σώμα και η ψυχή της Ευρώπης με συμμετοχή ε, σημαντικών προσωπικότητων από τον πολιτιστικό τομέα και ε, αυτή υποβλήθηκε τον τρίτο μήνα του 2014 με ένα από τα βασικά συμπεράσματα να είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά πράγματα. Αυτό με φέρνει τώρα στη δεύτερη φάση του αφηγήματο, δηλαδή τις προπαρασκευαστικές δράσεις τις οποίες εφαρμόζουμε τώρα και για τις οποίες θα σας ενημερώσω σήμερα. Πράγματι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι γνωρίζουμε τι αναμένουν οι πολίτες από την Ευρώπη αν αρκεστούμε μονάχα στα όσα συζητούνται εδώ στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό αποφασίσαμε να διευρύνουμε την συζήτηση ώστε να μπουν όλοι από τις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης. Εγώ θέλησα το project αυτό να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε ποια πράγματα μας ενώνουν, ποιε είναι οι κοινέ μας πολιτιστικές αξίες του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Θέλουμε να εξετάσουμε τις καθημερινές προτεραιότητες και τους αγώνες του ευρωπαίου πολίτη και να βρούμε μέσα από αυτές μια κοινή πολιτική αξία και το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η Ευρώπη. Εγώ ήθελα οι βασικοί ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι νέοι για το μέλλον της Ευρώπης, να βρεθούν στο επίκεντρο της συζητήσεως. Μερικοί λένε ότι οι νέοι απομακρύνονται από την πολιτική. Εγώ δεν έχω τέτοια εμπειρία. Η νεότερη γενεά έχει ξεκάθαρες απόψεις και θέλει να τις μοιραστεί με εμά. Ψάχνουν όμως να βρουν νέους τρόπους συμμετοχής στα κοινά πολλοί απομακρύνονται από τον τρόπο με τον οποίο δράει η πολιτική, γιατί θεωρεί ότι δεν λαμβάνει υπόψη τι ανησυχίε του. Χρειάζεται λοιπόν να γεφυρώσουμε το χάσμα γενναιών και να έρθουμε κοντά στου νέου. Για να γίνει αυτό πρέπει να φανούμε δημιουργικοί και να τους προσεγγίσουμε με τρόπους που να τους ενδιαφέρουν. Εκτός από, αυτού, οι νέοι, εκτός από αυτό οι νέοι έχουν δυναμισμό και δημιουργικότητα και αντιμετωπίζουν τα τρέχοντα προβλήματα της Ευρώπης με νέο τρόπο και με φρέσκια ματιά προσκάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο που μας πέρασε 7.000 νέες και νέους και οι ιδέες που κατέθεσαν είναι εντυπωσιακές και πραγματική έμπνευση για μας. Έχω περιλάβει λοιπόν στο project <clears throat> ορισμένες πτυχές. Στην πρώτη φάση διόρισα ε, μια ομάδα πρέσβεων για να συζητήσουν τα θέματα αυτά μέσα από τα διάφορα δίκτυα. Θέλω να τους ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς για την δέσμευση που έδειξαν και το πολύτιμο έργο που επετέλεσαν. Σήμερα θα σας εξηγήσουν τις απόψεις τους για το ευρωπαϊκό αφήγημα. Ε, ενσωματώσαμε επίσης οργανώσεις νέων και το European Youth Forum για να συζητήσουν πράγματα που οι νέοι θεωρούν σημαντικά. Τα μέλη επίσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ορισμένες από τις συζητήσεις αυτές. Για την παιδεία, για τα διάφορα δίκτυα του Erasmus ΣΥΝ, με συμμετοχή νέων από σχολεία, πανεπιστήμια, όλοι αυτοί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο νέο ευρωπαϊκό αφήγημα. Έχουμε και πολλά βίντεο όπου βλέπουμε τους νέους να μας εξηγούν ποιες είναι οι απόψεις τους για την ποικιλότητα στην Ευρώπη. Έχουμε περιλάβει και τους ασκουμένους στα ε, όργανα μας που έχουν, σε μοναδι... έχουν βρίσκονται στη μοναδική θέση να γνωρίζουν τα τεκτονόμενα στην Ευρώπη αλλά να τα βλέπουν μια φρέσκια ματιά. Θα δούμε το πρώτο βίντεο από τους ασκουμένους που παρήχθη τον προηγούμενο Φεβρουάριο και σε λίγες εβδομάδες όταν θα τελειώσει η φάση αυτή θα ε, δημοσιευτεί το επόμενο. Περιλαμβάνουμε στο νέο ευρωπαϊκό αφήγημα πολλές δραστηριότητες στον πολιτιστικό τομέα γιατί έτσι θα μεταφερθούν οι ιδέες και θα δώσουμε έμπνευση σε προβληματισμό και στοχασμό. Έχουμε τις αξίες που αποτελούν θεμέλιο της Ευρώπης και ε, τα θέματα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα, όπως θρησκείες κλπ, αλλά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε για να αντιμετωπίσουμε την ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Αυτό είναι από τις πιο σημαντικές και επίγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Είμαι πεισμένος ότι σημαντική θα είναι η προσφορά των ίδιων των νέων. Από το νέο ευρωπαϊκό αφήγημα των νέων μαθαίνουμε ήδη ότι αυτοί επιθυμούν μια Ευρώπη όπου η διαφορετικότητα θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση μιας κοινή ενισχυμένης ευρωπαϊκής ταυτότητας και όχι ενάντια σε αυτήν. Έχουμε αρχίσει λοιπόν τη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά δίκτυα νέων, τους οποίους θεωρούμε ανεκτήμητους εταίρους. Αλλά πού θα πάμε μετά. Τώρα συλλέγουμε ιδέες που μας προσφέρουν έμπνευση και προτάσεις που προέρχονται από τις διάφορες συζητήσεις και θέλουμε να μοιραστούμε με το υπόλοιπο της Ευρώπης. Άρχισα μόλις τώρα μια πλατφόρμα επιγραμμική διαβούλευσης που προσκαλώ τους νέους να ε, συμβάλλουν με τις ιδέες τους καθώς εξελίσσονται οι συζητήσεις. Για τέσσερις τομείς που προέκυψαν από τις συζητήσεις μας για το νέο ευρωπαϊκό αφήγημα ενωμένη στην πολυμορφία, απασχόληση και εκπαίδευση, ελευθερία διακίνησης και αλλαγή κλίματος. Στις αρχές του 2017 θα εξετάσουμε συλλογικά τα αποτελέσματα και θα διαμορφώσουμε το νέο ευρωπαϊκό αφήγημα σε ένα νέο, ε, νέο φορμά. Αυτό θα δείξει τι μπορούμε να κάνουμε μαζί για να προσφέρουμε ένα ρεαλιστικό όραμα σχετικά με τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε που είναι κατανοητό από όλες και όλους τους Ευρωπαίους και ιδίω να προσελκύσει τις νέες και τους νέους για να βοηθήσουν να φτιάξουμε την Ευρώπη του μέλλοντος. Θα χρησιμοποιήσω μάλιστα τα αποτελέσματα του νέου ευρωπαϊκού Αφηγήματο για να δώσω νέα όθηση στα ήδη υπάρχοντα βήματα όπως έρασμο συν, διαθωτικό διάλογος με τη νεολαία, ε, ε, διασκέψεις νέων, αθλητικά γεγονότα και επίσης chat, δηλαδή συζητήσεις διαδικτυακά. Έχω και άλλη σημαντική πρωτοβουλία για να ακούσουμε τις ιδέες και τις απόψεις ενός εκατομμυρίου νέων και επιγραμμικά και εκτός διαδικτύου μέχρι τέλους της θητείας μου. Στην Κόσιτσα τον Οκτώβρη θα κάνουμε ένα ακόμη βήμα και θα φτιάξουμε και την θα παρουσιάσουμε μάλλον τη διαδικτυακή πύλη. Πολύ συχνά ο διάλογός μας με τους νέους στρέφεται γύρω από τρέχουσες επικαιρότητες, ε, ε τρέχουσες, ε, τρέχουσα, τρέχοντα μάλλον επίκαιρα θέματα. Θα έχουμε όμως και άλλες δράσεις και θα δώσουν έμπνευση στην Κομισιόν για το πώς θα έλθει σε επαφή με τους πολίτες και πώς θα επικοινωνήσει με τους νέους και μέχρι τι επόμενε ευρωεκλογέ. Αυτό ενδιαφέρει πολύ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σα προσκαλέσω όλου και όλου να συμμετάσχετε στι συζητήσει στι χώρε μέλη, αλλά και τι επιγραμμικέ διαβουλεύσει. Εσεί παίζετε ένα σημαντικό ρόλο για να διαμορφώσετε συζητήσει στι οποίε συμμετέχουν και οι ψηφοφόροι σα. Και πολύ ευχαρίστω θα δεχθώ τι ιδέε σα για την τελευταία φάση τη προπαρασκευαστική δράσεω. Πριν ακούσω τώρα τι σκέψει σα, είμαι περίεργος να ακούσω και τις απόψεις ορισμένων εκ των πρεσβευτών μας για το νέο ή μάλλον για τα νέα ευρωπαϊκά αφηγήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι προτάσεις. Νομίζω ότι από πλευράς ε, Επιτροπής Πολιτισμού υπάρχει κάθε πρόταση να συνεισφέρουμε και να τροφοδοτήσουμε αυτή τη πλατφόρμα προγραμμάτων. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η ιδέα της συνάντησης που θα γίνει πριν από το 2017, μετά το καλοκαίρι δηλαδή, και η ιδέα μιας δικτυακής πύλης που θα συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να έχουμε και μαρτυρίες και σκέψεις των ε, πρεσβευτών μας, ε, των αξιότιμων προσκεκλημένων μας. Ε, θα μπορούσαμε να δώσουμε το λόγο στον καθένα ε, για πέντε λεπτά περίπου ή δυνατόν, να περιοριστείτε στα πέντε λεπτά. Πρώτα όμως θα δούμε το βίντεο. Νόμιζα ότι ήταν μετά. Πρώτα λοιπόν θα δούμε το ε, βίντεο και μετά θα δώσουμε το λόγο στους ομιλητές μας. Αν μπορούμε να κατεβάσουμε και λίγο το φωτισμό, να χαμηλώσουμε τα φώτα.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 trovo ε, molto Πολύ ενδιαφέρον αυτό το βίντεο. Συγχαρητήρια στο δημιουργό του. Ίσως θα μπορούσε να ε, κυκλοφορήσει και σε διάφορες γλώσσες για τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ε, και να αποτελέσει ένα μήνυμα για το τι θέλουν τα νέα παιδιά για την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό ότι του δώσαμε λίγο χώρο για να το εκφράσουν. Και τώρα θα ακούσουμε λοιπόν Ε, τους πρέσβεις μας και έχουμε παρουσία και των νέων. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Πάτρικ Κόβαξ, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΖΕΝ, της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Νέων Επιχειρηματιών. Παρακαλώ. We heard so many times that... Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι οι νέοι έχουν το κλειδί του μέλλοντος. Όμως, πόσες φορές τους ρωτήσαμε ποια πόρτα θέλουν να ανοίξουν με αυτό το κλειδί ή πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτό το κλειδί. Το νέο αφήγημα είναι ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για να το διαπιστώσουμε. Και το ότι καλέσαμε τόσους πολλούς νέους ανθρώπους να μας απαντήσουν με την πρωτοβουλία του Επιτρόπου, πιστεύω πως ε, είναι κάτι που θα μας βοηθήσει. Θα διεξαχθούν συνολικά 25 ε, συνέδρια γι' αυτό. 10 έχουν ήδη λάβει χώρα και τα υπόλοιπα 15 αναμένονται. Σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης, την ε, Γαλλία, την Πολωνία, την Τσεχία, το Βέλγιο και είναι όλα του σημαντικά. Αυτό που μας δίδαξαν οι νέοι είναι ότι χρειάζεται να αυξήσουμε την επικοινωνία και χρειάζεται να συνεχιστεί αυτή η επικοινωνία. Επειδή η επικοινωνία σημαίνει κατανόηση. Και η γενιά μας απαιτεί κατανόηση. υπάρχουν πολύ δραστήριοι νέοι άνθρωποι που ε, συμμετέχουν στα δρόμενα, είτε είναι μέλη οργανώσεων νεολαία, είτε, είτε οργανώσεων πολιτών, επιχειρηματιών. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που έχουν ενεργό ρόλο και θέλουν η φωνή τους να ακουστεί, οι οποίοι όμως ε, δεν είναι μόνοι. Θέλουμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και σε εκείνους που δεν είναι ενεργοί, που δεν είναι ε, προορατικοί. Γι' αυτό λοιπόν με μεγάλη μου χαρά βλέπω το πρόγραμμα αυτό, το νέο αφήγημα να επεκτείνεται και σε άλλα στρώματα και να συμπεριλαμβάνει λεώνα και περισσότερους νέους ανθρώπους οι οποίοι ε, δεν έχουν μόνο φυσική παρουσία αλλά και παρουσία στο διαδίκτυο και αν ακούσουμε και αφουγκραστούμε αυτούς τους νέους θα μάθουμε και τι ε, έχουν ανάγκη, τι θέλουν. Μετά από αυτά τα συνέδρια έχουμε αρκετά ευρήματα. Όπως είπε και ο κύριος Ναύρατσιτς, οι νέοι θέλουν να συμμετέχουν. Υπήρχε μάλιστα και μία συζήτηση για να μειωθεί η ηλικία όπου μπορεί κάποιος να ψηφίσει από τα 18 στα 16. Τους νέους επίσης τους απασχολεί το μεταναστευτικό ζήτημα και η ένταξη των μεταναστών. Θέλουν περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερη πρόσβαση που να γίνεται και μέσω των ε, κοινωνικών μέσων. Πολλέ φορές στα μέσα ενημέρωση διαβάζουμε ότι στις Βρυξέλλες λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις και οι νέοι λοιπόν θέλουν να συναντήσουν εκείνου που λαμβάνουν τις αποφάσεις και να έχουν μία σωστή και δίκαια επικοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε πως το νέο φύγημα για την Ευρώπη είναι η σωστή πλατφόρμα γι' αυτό. Οι νέοι όμω θέλουν και να ζουν σε μία Ευρώπη η οποία δεν θα φοβάται τα λάθη το 1 τρίτο των νέων στην Ευρώπη θέλει να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα σε ε, αντιδιαστολή με το 2 τρίτα των νέων στην Ασία. Και αυτό γίνεται ε, διότι υπάρχει φόβος αποτυχίας. Οι νέοι θέλουν να μάθουν, θέλουν να χτίσουν γέφυρες ε, ανάμεσα στις γενιές και ανάμεσα στα έθνη. Γι' αυτό λοιπόν μπορώ να πω πολύ περήφανα ότι η δική μας γενιά θέλει να μάθει, θέλει να ακούσει, είναι ανοιχτή, αλλά πάνω απ' όλα εκτιμά την ευκαιρία να εκφραστεί και να της δείξουν την πόρτα στην οποία, την οποία θέλουν να ανοίξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την μαρτυρία σας. Ε, είναι και εξ ονόματος ε, νέων επιχειρηματιών, επομένως είναι πολύ ενδιαφέρον για μας ε, να σας ακούμε. Και τώρα ο λόγος του Μίκαλ Κλάιμπερ, ερευνητή και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Επιστημών της Πολωνίας. Επιτρέψτε μου να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι θεωρώ τιμή μου το γεγονός ότι συμμετείχα σε αυτή την πρωτοβουλία εδώ και κάποια χρόνια, διότι μου προσφέρει την ευκαιρία να προωθήσω την ιδέα της κοινή Ευρώπης. Μια ιδέα που ε, αγαπώ ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι αγαπά και η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων. Σίγουρα συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους ε, απόψεις των οποίων συνόψισε ο Επίτροπος, αλλά θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία τα οποία αφορούν την προσωπική μου εμπειρία. Καταρχάς, Προσυπογράφω τα όσα είπε ο συνάδελφος προηγουμένως. Η νέα γενιά είναι αυτή η οποία πρέπει να έχουμε κατά νου για να παρουσιάσουμε το μέλλον της Ευρώπης με ελκυστικό τρόπο, διότι η νέα γενιά είναι αυτή η οποία θα ζήσει στην Ευρώπη και είναι αυτή η νέα γενιά η οποία θα υποφοληθεί από τη ζωή στην Ενωμένη Ευρώπη. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας στο μέλλον. Η δεύτερη παρατήρησή μου, η οποία βασίζεται φυσικά και στην εμπειρία μου, είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στον τρόπο με τον οποίο συζητούμε για το μέλλον της Ευρώπης και όχι ιδεαλιστές και αφελείς. Αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό και στη συζήτηση στην οποία συμμετείχα άκουσα πολλές εμπειρίες που έλεγαν ότι μπορούμε να επικαλιστούμε αρκετά επιχειρήματα υπέρ του μέλλοντος της Ευρώπης που είναι ρεαλιστικά και γίνονται πολύ καλύτερα αποδεκτά τη σήμερον ημέρα στον περίπλοκο κόσμο στον οποίο ζούμε. Τρίτο σχόλιο. Εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, επομένως το φυσικό μου περιβάλλον είναι ο πανεπιστημιακός κόσμος ερευνητές και φοιτητές δηλαδή. Και καταρχάς θεωρώ ότι η έρευνα και η ανώτατη εκπαίδευση είναι σαφώς αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού. Και δεύτερον, οι ομάδες αυτές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα ε, όταν τους μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης, διότι οι ερευνητές εξορισμού ε, έχουν ε, ένα μυαλό διεθνέ. Δεν μπορεί να κάνει έρευνα στο σπίτι σου, πρέπει να συνεργαστεί. Και η άλλη ομάδα, οι φοιτητέ, κατά την άποψή μου, και το πιστεύω ακράδαντα αυτό, είναι ε, μια ομάδα που είναι ο μεγαλύτερος υπέρμαχος της Ευρώπης σε σχέση με τους υπολείπους. Όταν συζητώ με φοιτητές σε πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη, έχω την αίσθηση ότι πραγματικά ζω σε μία Ευρώπη. Χάρη και στα προγράμματα ανταλλαγή ε, και σε άλλες πρωτοβουλίες, έχουμε ε, ένα διεθνές ακροατήριο όποτε μιλούμε ε, στο Πανεπιστήμιο και αυτό δημιουργεί προσδοκίες να αλλάξουμε τα πράγματα στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι ε, που αναπτύσσεται αυτό το πνεύμα. Τελευταίο σχόλιο. Η ομάδα αυτή που σας ανέφερα είναι αυτομάτως υπέρμαχοι της Ευρώπης ε, στην οτροπία τους, αλλά πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να μιλήσουν. Διότι αφήνουμε αυτές τις φωνές ε, στη συζήτηση για την Ευρώπη και τις παραμελούμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έκανα μια παρουσίαση για να προσπαθήσω να παρουσιάσω αυτό το νέο αφήγημα για την Ευρώπη σε 120 ε, άτομα στο Σάλτσπουργκ στην Αυστρία και ήταν ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό συνέδριο και το αποτέλεσμα ήταν ότι κατάφερα να ξεκινήσω ένα πρόγραμμα με τον τίτλο Next Europe, η επόμενη Ευρώπη, που περιλαμβάνει τώρα εκατοντάδες ερευνητές ανά την Ευρώπη, σε μία απόπειρα να διαμορφώσουν και να βοηθήσουν να εκφραστούν ιδέες οι οποίες θα βοηθήσουν αυτό το νέο φύγημα για την Ευρώπη. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε στις ομάδες των νέων ανθρώπων και πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να μιλήσουν, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πεπισμένοι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο να συμπορευτούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για αυτή τη μαρτυρία σας και για το γεγονός ότι πολύ σωστά επικεντρώνεστε σε αυτές τις δύο ομάδες ε, ανθρώπων που είναι εκφύσεως περισσότερο ευρωπαϊστές και θα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση, θα έπρεπε μάλλον να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση ε, για να μιλήσουν. Να δώσουν τώρα το λόγο στην κυρία Σνέσκα Κουάτλεκ Μιχαήλοβιτς, ε, Γενική Γραμματέα του, ε, της δικής μας Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ <clears throat> κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας θυμήσατε ότι σήμερα είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Και ο πρόεδρος μου, ο ε, τενόρος Πλάση του Ντομίνγκο, θα είναι πολύ χαρούμενος που σήμερα συζητεί το Ευρωκοινοβούλιο το νέο ευρωπαϊκό αφήγημα, διότι ο στόχος όλου αυτού του εγχείρηματο είναι αυτή η μετακίνηση του τρόπου με, τον οποίο μιλούμε για την Ευρώπη, αντιλαμβανόμαστε την Ευρώπη, αυτή η πραγματική αλλαγή του τρόπου, όπω λέω που μιλούμε για την Ευρώπη, αντί πλέον με οικονομικού όρου να μιλήσουμε με όρου πολιτισμού. Κάτι το οποίο θα μα βοηθήσει ασφαλώ να αναζωογονήσουμε αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα και ας τολμήσω να το πω, να κάνουμε και τους Ευρωπαίους πολίτες, τις νέες και τους νέους, να αγαπήσουν ξανά την Ευρώπη. Θεώρησα λοιπόν μέγα προνόμιο για μένα που ήμουν από τις πρώτες που συμμετέσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Επίτροπο Ναύρατσης που με διόρισε μαζί με τους άλλους συναδέλφους μου εδώ ως πρέσβυρα σε αυτή τη δεύτερη φάση. Δεύτερη φάση που νομίζω αγαπητέ Επίτροπε ότι σωστά επιλέξατε να βάλετε άλλη μια κίνηση, να ρίξετε δηλαδή το βάρος, να ε, ε, φέρετε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την νεολαία. Μπορείτε, δηλαδή, μπορέσατε δηλαδή με τις προσπάθειές σας να φέρεται να συμμετάσχουν όλες οι οργανώσεις νεολαίων. Κάτι το οποίο έλειπε από την πρώτη φάση. Έχουμε φτιάξει λοιπόν αυτό το μεγάλο δίκτυο τώρα στην δεύτερη φάση. Δικός μου ρόλος ως πρέσβυρας του νέου ευρωπαϊκού αφηγήματος είναι να πω ότι ελπίζω ότι θα υπάρξει και μια τρίτη και τελική φάση του εγχειρήματο που θα αποτελέσει την σύνθεση εν τέλει, που θα μας επιτρέψει δηλαδή να φέρουμε κοντά όλες αυτές οι πρωτοβουλίες τα άτομα, τους νέους, τις νέες, τους επιστήμονες, τους καλλιτέχνες, την πολιτιστική κληρονομιά, να τους φέρουμε να προσεγγίσουν δηλαδή. Και εμείς θα θέλαμε να υπάρξουν πολύ περισσότερες γέφυρες μεταξύ των θαυμάσιων πρωτοβουλειών στον χώρο του πολιτισμού, της παιδείας και βεβαίως οτιδήποτε έχει να κάνει με τους νέους. Επειδή είμαι και γενική γραμματεύς της Ευρώπα Νόστρα, που είναι η φωνή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, χρησιμοποιώ την ευκαιρία για να δηλώσω ότι επιθυμώ το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς που είναι το 2018 και να ευχαριστήσω βεβαίως το Ευρωκοινοβούλιο που τόσο πολύ υποστήριξε όλες και όλοι σας αυτή την πρωτοβουλία. Να πω λοιπόν ότι πρόκειται για μια θαυμάσια πρωτοβουλία για να προωθήσουμε αυτό το νέο ευρωπαϊκό αφήγημα το οποίο είναι νέο αλλά είναι και βασισμένο ταυτόχρονα στην κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία. Δεν μπορούμε να γράψουμε νέα κεφάλαια του βιβλίου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας εάν δεν γνωρίζουμε τα προηγούμενα, από πού ήρθαμε δηλαδή και ποιες είναι οι κοινέ μας αξίες. Έτσι λοιπόν το 2017 ελπίζω το νέο ευρωπαϊκό αφήγημα θα συμβάλλει ώστε να φτιάξουμε αυτή τη γέφυρα. Και βεβαίω και η πολιτιστική διπλωματία, άλλη σημαντική δραστηριότητα. Και αυτή προστίθεται στο, προστίθεται στο νέο ευρωπαϊκό αφήγημα και δίνει την έμφαση σε αυτή την ήπια δύναμη που είναι η Ευρώπη εγώ πιστεύω ότι αυτό το sharing, ακούσαμε και στο, και στο βίντεο, sharing and caring, δηλαδή να τα μοιραζόμαστε όλα και να φροντίζουμε ένα στον άλλο. Και η, το μοίρασμα αυτό της κοινή κληρονομιάς είναι επίσης το ίδιο σημαντικό. Και για να επανέλθω στην μουσική, μόλις προ τριών εβδομάδων ο Επίτροπος Ναυρατσίτς μαζί με τον πρόεδρό μου, τον μαέστρο ε, Πλάσιο Ντομίνγκο στην θα θέλω στη Μαδρίτη γιορτάσαμε την απόφαση και τα βραβεία της Ευρώπα Νόστρα για να γιορτάσουμε την κοινή μας χρονομιά και μέσα στην Ευρώπη αλλά και μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Αυτό είναι το μήνυμά μου, στο οποίο πιστεύω απόλυτα και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το συνοδεύω με την ευχή ότι θα μας υποστηρίξετε και στην τελευταία αυτή φάση, αλλά ότι θα συμμετάσχετε κιόλα όλε και όλοι. Διότι θέλουμε να μας στηρίξει χρηματοδοτικά το Κοινοβούλιο, το χρειαζόμαστε αυτό, αλλά θέλουμε και την δική σας προσωπική συμμετοχή. Και γιατί όχι, να κάνετε και μια συζήτηση και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το νέο ευρωπαϊκό αφήγημα. Χρειαζόμαστε την προσπάθεια όλων των Ευρωβουλευτών. Και η τελευταία αυτή διασύνδεση θέλω να κάνω μεταξύ πολιτισμού, νεολαία και βεβαίω του ανώτατου αυτού επίπεδου εκπροσώπησης των λαών και τοπικού και ευρωπαϊκού βεβαίω. Ευχαριστώ πολύ και για τον ενθουσιασμό σας που ποτέ δεν μας λείπει. Και φυσικά και για αυτές τις τελευταίες σας προτάσεις, ε, οι οποίες αξίζουν να τις ε, μελετήσουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Η ιδέα είναι να έχουμε μια πιο πολιτιστική ε, χρειά στην Ευρώπη, επομένως είναι και ε, ε, κεντρική σημασία το θέμα αυτό εν ώψη και του 2018. Και τώρα ο λόγος στον Πολ του Ζαρντάν, τον οποίο σα παρουσίασα προηγουμένω, διευθυντή ε, του κέντρου Μποζάρ των καλών τεχνών στι Βεξέλλε, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν εκ των πρωταγωνιστών στο θέμα αυτό. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητέ Επίτροπε, Θα συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφός μου. Πιστεύω ότι το ερώτημα εδώ είναι κάτι που πρέπει να αφορά όλους, όλα τα θεσμικά όργανα. Ακόμα και τους επόμενους μήνες θα πρέπει να μας απασχολήσει έτσι ώστε να βρούμε λύση, διότι ακόμα και αν λείπουν οι υπόλοιποι πρέσβεις, θα ήθελα και εγώ να μιλήσω εκ μέρους σε κάποιων καλλιτεχνών. Είμαστε εκπρόσωποι όλων που συμμετέχουν σε αυτό το project. Και θα έλεγα ότι εδώ είμαστε στο πρώτο στάδιο της προσπάθειας και ελπίζω σε επόμενο στάδιο οι καλλιτέχνες ε, και οι νέοι άνθρωποι να καθίσουν μαζί με τους πολιτικούς για να ανταλλάξουν απόψεις. Ε, διανοούμενοι πολιτικοί καλλιτέχνες μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ως κομμάτι αυτού του αφηγήματο να χτίσουμε γέφυρες με συγκεκριμένο τρόπο. Επιπλέον, στη, στο Μποζάρ μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίσαμε ένα project όπου προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με την επόμενη γενιά. Το πώς δηλαδή θα χτίσουμε γέφυρες ανάμεσα στον κόσμο της τέχνης, ε, ανάμεσα στα σχολεία, στον κόσμο των επιστημών και στον κόσμο των επιστημών. Καταλήξαμε στο να συνεργαστούμε με πάνω από 100.000 μαθητές στο Βέλγιο, διότι Πιστεύουμε σε αυτούς και πιστεύουμε και στις αξίες της Ευρώπης. Η γνώση λοιπόν και οι αξίες. Προσπαθήσαμε να συνδέσουμε αυτά τα δύο πάνω σε αυτό το project στο οποίο συμμετείχαν νέοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι κλήθηκαν να μεταφράσουν τις ιδέες και τις ελπίδες τους σε εικόνες. Το πώς δηλαδή θα χτίσουν γέφυρες. Ο Επίτροπος ήθελε εκπαίδευση, ήθελε ε, να ασχοληθεί με την νεολαία και εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε γέφυρες ανάμεσα στα, ε, στο πρώτο project και στα επόμενα. Να δημιουργήσουμε μία συνέχεια δηλαδή ανάμεσα στην, ε, στο Creative Europe και στα άλλα project που θα έρθουν. Να τα συνδέσουμε με διάφορα άλλα προγράμματα της Επιτροπής όπως το ψηφιακό θεματολόγιο ελπίζω τους ερχόμενους μήνες με την ιδιότητά μου ως πρεσβευτής να βοηθήσω έτσι ώστε να πληροφορηθούν όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι για αυτά τα προγράμματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα αφηγήματα να γίνουν γνωστά και εντός και εκτός Ευρώπης. Μην ξεχνάτε ότι αυτό ε, είναι η πολιτισμική διπλωματία που ακούμε και ότι οι χώρες που βρίσκονται στη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμπεριληφθούν και πρέπει να μάθουν για αυτές τις ε, αξίες. Πρέπει λοιπόν να διαδοθούν και εντός και εκτός Ευρώπης. Ε, να μιλήσουμε για τη μετανάστευση, για τη διαφθορά, για το κοινωνικό ντάμπινγκ. Και εάν δυσκολεύονται οι πολιτικοί, δυσκολεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε τη σκητάλη μπορούν να την αναλάβουν οι καλλιτέχνε οι οποίοι θα μεταδώσουν αυτέ ε, τι αξίε. μέσω ε, του πολιτισμού, μέσω της τηλεόρασης, των ε, σειρών για παράδειγμα. Να δούμε δηλαδή και εκεί για το πώς ε, θα δημιουργήσουμε αυτό το αφήγημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε και από τον Πόλτιο Σαντεντάν Πριν δώσω το λόγο ε, στους συναδέλφους, να δώσουμε για ένα λεπτό το λόγο στον κύριο Λόκεγκαρτ, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής αυτής της πρωτοβουλίας το 2013 και ακόμα την παρακολουθεί και μετά θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Παρακαλώ κύριε Λόκεγκαρτ. Θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Ένα λεπτάκι μόνο. Και ευχαριστούμε και για την παρουσία σας εδώ. ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω λίγα πράγματα πάνω σε αυτά που ήδη υπόθηκαν. Να ευχαριστήσω καταρχάς τους πρέσβεις και τον κύριο Επίτροπο που ήρθαν εδώ. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η ιδέα του να γεφυρώσουμε δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς ως πολιτικοί με άλλους τομείς, με τις επιστήμες, με τον πολιτισμό, με την εκπαίδευση, με την νεολαία, είναι κατά τη γνώμη μου το κλειδί για όλο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Το σκεπτικό πίσω από αυτό το εγχείρημα ήταν ακριβώς αυτή η δημιουργία ε, συνδέσεων. Ακριβώς το να χτίσουμε αυτές τις γέφυρες. Ανάμεσα στους πολιτικούς και στους υπόλοιπους, στους μη πολιτικούς. Και είναι κάτι που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Γι' αυτό και εγώ στηρίζω αυτή την ιδέα, γιατί πιστεύω πως έτσι θα πάμε μπροστά. Και αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Επίτροπε που αναλάβατε αυτήν την πρωτοβουλία, διότι χρειαζόμαστε και πολιτισμό και τις επιστήμες και τους νέους για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες μας για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα διότι ας παραδεχτούμε πως εμείς ε, οι πολιτικοί έχουμε αποτύχει και πρέπει να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών και αυτό θα το κάνουμε παίρνοντα με το μέρος μας τις ε, επιστήμες, τον πολιτισμό, τους νέους. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να συμπεριλάβετε αυτές τις γέφυρες στο μελλοντικό σας πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι και είμαι βέβαιη ότι αυτή η γέφυρα θα πρέπει να παραμείνει. Δηλαδή, πρωτοτυπία του νέου φυγήματος, αλλά και ταυτόχρονα ε, το, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προσδώσουμε και μια πολιτική διάσταση στο θέμα, γιατί αυτή είναι υποχρέωση όλων. Το λέμε εμείς ε, συνέχεια ως πολιτικοί, ως ευρωβουλευτές, ότι ορισμένες φορές δίνεται η εντύπωση ότι σε αυτές τις στιγμές, τις τόσο σημαντικές που ζούμε, υπάρχει απόλυτη ανάγκη να γίνεται ένας ανοιχτός, μόνιμος, επικριτικός διάλογος με τον κόσμο του πολιτισμού, τις έρευνες των σχολείων, των πανεπιστημίων, με ε, μόνιμη παρουσία των νέων και νεών, χωρίς όμως να χάνουμε και αυτή τη διάσταση του διαλόγου που χρειαζόμαστε ε, εκατέρωθεν νομίζω. Τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Η κυρία Ζωηντρόβα πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους πρέσβεις που ανέπτυξαν τα θέματα. Είναι σημαντική η εμπειρία αυτή και για μας. Θα επανέλθω σε κάτι που είπε ο Μιχάλ Κλάιμπερ, ότι η σπουδαστές είναι η πιο ενσωματωμένη ομάδα για, τους, για την Ευρώπη. Η πιο δηλαδή δεσμευμένη και διότι οι σπουδαστές είναι υπέρ της Ενωμένη Ευρώπης και συμφωνώ και συμφωνώ με αυτούς διότι πολλοί θεωρούν την ελεύθερη Ευρώπη σαν κάτι τόσο αυτονόητο που δεν θεωρούν ότι χρειάζεται να κάνουν καμία προσπάθεια για να την διατηρήσουν. Γι' αυτό χρειάζονται και τις εμπειρίες των γονιών τους. Οι συνέπειες που βλέπουμε σήμερα είναι ότι ο εξτρεμισμός κερδίζει έδαφος και από αριστερά και από δεξιά. Είναι σημαντική η παρουσίαση του προγράμματος για το νέο ευρωπαϊκό αφήγημα. Έχουν σημασία όμως οι προσωπικότητες. Οι απόψεις σημαντικών προσωπικότητων που να λάβουν το λόγο και να μιλήσουν στους νέους, στις νέες, στους πολίτες. Και στο έργο, στο project αυτό που έχετε προτείνει, βλέπω ότι λαμβάνουν το λόγο και άνθρωποι και από την πολιτική ζωή και από την επιστήμη και από την παιδεία Τώρα κοιτάξτε, είμαστε δύο μέρες πριν από το Βρετανικό δημοψήφισμα. Είμαι βεβαία ότι εάν κάτι μπορεί να επηρεάσει τους Βρετανούς να καταψηφίσουν το Brexit, δεν θα είναι τα λόγια του Πρωθυπουργού Κάμερον. Αλλά θα είναι πιο πολύ η θυσία των εισαγωγικών της βουλευτού Τζοε Κόξ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για αυτή την αναφορά, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ε, Εχθέ στην έναρξη της συνεδριασής μας αποτίσαμε φόρο τιμής ε, στη μνήμη μια γυναίκας η οποία πλήρωσε με τη ζωή τη ε, την αγάπη τη για την Ευρώπη εν τέλει. Η κυρία Λιμπάτσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. <clears throat> Άκουσα και τον Επίτροπο και τους προσκεκλημένους. Όταν μιλούμε για την μελλοντική πορεία της Ευρώπης και αν θέλουμε ένα νέο ευρωπαϊκό αφήγημα, πρέπει πρώτα να θέσουμε σε αυτούς το ερώτημα ποια είναι τα φυσικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και όταν υπήρχε ακόμη το σίδηρον παραπέτασμα, υπήρχε ωστόσο μια κοινότητα πολιτισμού και μια κοινότητα επιστήμης και γνώσης. Η συνεργασία στην Ευρώπη αναδείχνονταν ανεξάρτητα από τις πολιτικές δυσχέρειες. Τώρα, καλούμεθα να αναρωτηθούμε ποιος θα είναι ο ρόλος του πολιτισμού και της επιστήμης στην Ευρώπη και ποιο ρόλο θα παίξει η Ευρώπη για την ανάπτυξη της επιστήμης. Συμφωνώ με τον Επίτροπο Ναβρατσίτς ότι οι σημαντικότεροι αποδέκτες των προγραμμάτων και του νέου ευρωπαϊκού αφηγήματος θα πρέπει να είναι η, νέα, η νεολαία, συγγνώμη, διότι αυτοί οι νέοι, οι νέοι δηλαδή και οι νέες που θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον της Ευρώπης σε λίγα χρόνια. Όμως έχω να θέσω και ένα ερώτημα. Τι γίνεται τώρα. Στην εκπαίδευση βλέπουμε τους νέους και τις νέες να, γίνονται, να είναι φιλοευρωπαίοι. Μετά ριζοσπαστικοποιούνται όμως αργότερα. Υπάρχουν δηλαδή ε, ε, νέοι και νέες φοιτητές και φοιτήτρες που παραμένουν φιλοευρωπαίοι, αλλά άλλοι ριζοσπαστικοποιούνται. Εγώ θεωρώ ότι αυτά προκύπτουν από τις πρώτες εμπειρίες των νέων, στις πρώτες επαφές δηλαδή με τον επαγγελματικό κόσμο, με τον κόσμο του επαγγέλματος. Γι' αυτό και θέλω να ζητήσω, να πω το εξής, ότι αν θέλουμε νέο ευρωπαϊκό αφήγημα, θα πρέπει να διαμορφώσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία να συνδέουν και όχι να χωρίζουν τον κόσμο. Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια να μπορούν να συμμετέχουν όλες οι κοινωνικές ομάδες στα προγράμματα αυτά. Ανεξαρτήτως κριτηρίων. Παράδειγμα, όταν μιλήσαμε για το πρόγραμμα Έρασμος, είπαμε ότι διαπιστώσαμε δηλαδή ότι κοινωνικά μη προνομίχες ομάδες δεν είχαν επαρκή πρόσβαση το πρόγραμμα για το 2020, η Πολωνία έχει ένα σημαντικότατο ε, διανοητικό δυναμικό. Όμως η χρήση των ε, γνώσεων του δυναμικού αυτού είναι πάρα παραπολιτική. Έρχομαι στο σχέδιο Juncker. Πώς διαμορφώνονται τα έργα που ε, ενισχύονται από το πρόγραμμα αυτό. Πολλά είναι στην παλαιά Ευρώπη, πολύ λίγα είναι στη Νέα Ευρώπη, στο ανατολικό τμήμα της Ευρώπης δηλαδή. Εγώ χαίρομαι για το πρόγραμμα αυτό, αλλά να μην δυσμονήσουμε τα θεμέλια που είναι αυτά στα οποία βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε την Κριστίνα για αυτή την παθιασμένη παρέμβαση και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Στρογεύσκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Συμμετέχω εδώ και πολλά χρόνια σε αυτές τις συζητήσεις όπου συζητάμε για το πώς να ορίσουμε την Ευρώπη, ποια, ε, ποιο θα είναι το μελλοντικό αφήγημα για αυτή κτλ. Και κάθε μέρα που περνάει γίνομαι και πιο απεσιόδοξος, με κάθε συνάντηση ακόμα περισσότερο. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο αφήγημα. Δεν ξέρω αν αξίζει να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είναι αναγκαίο ένα νέο φύγημα, διότι φυσικά και είναι αναγκαίο. Όμως κάνουμε λάθη και το πρώτο ε, λάθος που κάνουμε είναι να αναρωτιόμαστε γιατί ε, πρέπει να υπάρχει ένα νέο αφήγημα, που θα ωφελήσει. Είναι σαφές, ε, πιστεύω, ε, το ότι πρέπει να υπάρξει ένα νέο αφήγημα. Όμως οι απόψεις δίστανται σχετικά με το ποιου, ποιους στόχους πρέπει να έχει και μία άλλη παρατήρηση. Φυσικά και καταλαβαίνω ότι το αφήγημα πρέπει να απευθυνθεί στους νέους. Ε, όμως το αν πρέπει να απευθυνθεί μόνο σε νέους ε, θα απαντούσα ναι υπό προϋποθέσεις όμως. Υπό την προϋπόθεση η Ευρώπη να μην ξεχάσει και τους ε, ηλικιωμένους. Η Ευρώπη πρέπει να κατανοήσει ότι χρειάζεται σεβασμός προς τους ηλικιωμένου και τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά τους. Ας δούμε το παράδειγμα, το υπόδειγμα θα έλεγα της Ιαπωνίας, όπου οι ηλικιωμένοι ε, απολαμβάνουν πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό και θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτό το καλό παράδειγμα. Ε, τώρα, ε, να πω ότι ανεξάρτητα με το τι θα γίνει ή όχι στο Βρετανικό Δημοψήφισμα την Πέμπτη, Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Έχουμε τον αθλητισμό, έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδροσφαίρου στην Γαλλία που πρέπει να το γιορτάσουμε. Όμως ε, ταυτόχρονα και το, την τραγωδία που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη δολοφονία της ε, βουλευτή η οποία πολεμούσε για ε, τα δικαιώματα στην πολυμορφία. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτήν την πολυμορφία, αυτήν την πρωτοτυπία. Από την άλλη όμως πρέπει και να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουν όλα αυτά στην Ευρώπη. Τι επιπτώσεις θα έχει στη νέα γενιά. Πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει στο μέλλον. Ο θα δούμε καλύτερους ζωγράφους από τον Van Gogh, τον Νταβίντσι, τον Μονέ, καλύτερους συνθέτες από τον Μπετόβεν, καλύτερους σκηνοθέτες από τον Μπέργκμαν και τον Βισκόντι. Να τονίσω κάτι. Ο πολιτισμός είναι ο σημαντικότερος ε, τομέας για επενδύσεις, για μελλοντικές επενδύσεις. Η Ευρώπη χρειάζεται νέες επενδύσεις, νέο περιεχόμενο. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ευρωπαϊκή πολιτική να ασχοληθεί με τον πολιτισμό και με τις επιστήμες. Είναι κάτι το, στο οποίο δεν δίνεται αρκετή προσοχή μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ απόλυτα με αυτή την τελευταία παρατήρηση και ελπίζω να είμαστε όλοι στην ίδια άγουσα. Θέλουμε δηλαδή του χρόνου στον προπολογισμό, μια και αναφερθήκατε στον προπολογισμό, να ληφθούν περισσότερο υπόψη τα προγράμματα για τον πολιτισμό. Η κυρία Κίνη Μπαρμπάτ τώρα έχει το λόγο. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ε, αξιότιμοι κύριοι Επίτροπε, αξιότιμοι ομιλητές που ήρθατε να μιλήσετε εδώ μαζί μας σήμερα για το ευρωπαϊκό αφήγημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον συνάδελφο Λόκεγκαρ για τα όσα κάνει και για την ε, δέσμευσή του για το έργο αυτό, το οποίο το θεωρώ πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τελείως διαφορετική εικόνα αναχώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, οι ε, στατιστικές δείχνουν ότι οι αρνητικές απόψεις κυριαρχούν και φαίνεται να υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση για την Ευρώπη. Για να το αλλάξουμε αυτό χρειαζόμαστε ένα αφήγημα το οποίο να είναι αξιόπιστο για την Ευρώπη και θα βασίζεται σε ισχυρές ιδέες, εύκολα αναγνωρίσιμες και κοινέ. Και θα ήθελα να σταθώ σε τρεις πυλώνες που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για αυτό το αφήγημα. Το πρώτο είναι ε, το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό μέλλον δεν είναι γραμμένο ε, είναι στα χέρια μας το να οικοδομήσουμε ή να καταστρέψουμε στην Ευρώπη. Δηλαδή η μελλοντική Ευρώπη, μελλοντικη ευρωπη της ευημερία δεν θα επιτευχθεί χωρίς προσπάθειες. Χρειαζόμαστε ε, βούληση και ευφυΐα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι μια αρχή του Ζαν Μονέ. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ένα σύνολο ανθρώπων ε, και όχι μια ένωση κρατών ή εθνών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινωνία η οποία θα βασίζεται στα ατομικά δικαιώματα, θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, με την απαραίτητη αξία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους ανταγωνιστές τους που είναι ε, πάρα πολλοί. Ο τρίτος πυλώνας είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο οικονομία. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι μια κοινότητα ανθρώπων, ε, πολιτισμών και αξιών οι άνθρωποι, αντίστοιχα με ό,τι λέγεται, δεν ανταποκρίνονται μόνο σε οικονομικά κίνητρα ε, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν πολλούνται. Οι θεμελιώδεις αξίες ε, τις οποίες πρέπει να υπερασπιστούμε και αυτές είναι η προσωπικότητα και η ουσία μιας πραγματικής κοινότητας. Ως εισηγήτρια της ε, εκτελεστικής έκθεσης ε, του προγράμματος «Μια Ευρώπη για τους πολίτες» θεωρώ ότι το έργο αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να συμπεριληφθεί σε αυτό το πρόγραμμα και να λάβει την κατάλληλη όθηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ τη συνάδελφο. Η κυρία Μπίλντε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καταλαβαίνει ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεσμικών οργάνων και Ευρωπαίων πολιτών και κυρίως των νέων ένα 27,8% ε, νέων 18 με 25 ετών ψήφισαν στις τελευταίες ευρωεκλογέ. Γεγονός που ε, αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής από το 1979. Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν χώρες οι οποίες πλήττονται με τεράστιο ποσοστό ανεργίας. Υπάρχουν ένα 22% ανέργων στην Ευρωζώνη και ένα 40% στο σύνολο της Ευρώπης. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τι χάσμα υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτών. Η λύση είναι τα βασικά εκτελεστικά όργανα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σεβαστούν καλύτερα τη λαϊκή βούληση και ίσω έτσι ε, θα είχαμε μια συμφιλίωση με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάβασα με προσοχή το σημείωμα το οποίο μας διαβιβάσατε για αυτό το νέο αφήγημα για την Ευρώπη και θα ήθελα να με διευκρινίσετε ότι αν λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει συζητήσεις, βίντεο, θετικά μηνύματα, ε, μπορείτε να μου πείτε πόσο στήχησαν όλα αυτά πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το νέο αφήγημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βερχάγεν. Χαίρομαι πολύ που βλέπω να αναπτύσσονται πολλές νέες ιδέες για την Ευρώπη, για τη νέα γενιά, που μπορούν να φέρουν αυτή λοιπόν τη νέα γενιά πιο κοντά στην Ευρώπη και την Ευρώπη πιο κοντά στους νέους. Όμως, αναρωτιέμαι πώς θα φτάσουμε στην πλειοψηφία των νέων, στην πλειοψηφία των πολιτών. Πώς θα το κάνουμε με φυλάδια, με εντό εισαγωγικών νέα αφηγήματα ή μήπως πρέπει να έρθουμε πιο κοντά στους ε, νέους, στους πολίτες μας με τις αποφάσεις που λαμβάνουμε, με την συμπερίληψή τους σε αυτές. Πώς θα γίνει αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες. Πιστεύω πως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα εφιστάμενα προγράμματα που ε, έχουμε στη διάθεσή μας, που τρέχουν, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς, έτσι, ώστε, ώστε να ενισχύσουμε την πληροφόρηση στα σχολεία, στα ε, διάφορα ε, δημόσια κτίρια. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να γίνει υποχρεωτικό μάθημα τα ευρωπαϊκά θέματα στα σχολεία. Πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον και πρέπει να προσπαθήσουμε να φέρουμε λοιπόν την Ευρώπη πιο κοντά στα σχολεία. Έτσι ώστε οι νέοι να έρθουν ε, σε αντιπαράθεση με την Ευρώπη, να έχουν μια πρώτη γνωριμία ήδη από τα σχολικά τους χρόνια. Πρέπει να φτιάξουμε μια Ευρώπη για τους πολίτες μας ξανά διότι πιστεύω πως αυτό είναι αναγκαίο και πρέπει μάλιστα να γίνει ε, νωρίς. Ε, το Εράσμους, το Λεωνάρντο, το Εράσμους Πλάς, το Κομένιος, αυτά τα προγράμματα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για τους πολίτες, για να έρθουμε πιο κοντά σε αυτούς. Διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μεγαλώσουμε μαζί και να ενηλικιωθούμε. Πιστεύω πω αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετέ εθνικιστικές τάσει που συναντάμε σε πάρα πολλέ χώρε τη Ευρώπη, τι οποίε πρέπει να καταπολεμήσουμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουν οι πολίτε για ποιο λόγο υπάρχει η Ευρώπη, για ποιο λόγο πρέπει η Ευρώπη να είναι ενωμένη. Δεν πρέπει να ξεχάσουν τι σημαίνει η ειρήνη, τι σημαίνει η διασυνοριακή συνεργασία. Αυτή τη στιγμή το ξεχνάμε. Γι' αυτό ε, οδηγούμαστε ε, στο να υπάρχει κίνδυνος να ξανακλείσουν τα σύνορα, να χάσουμε αυτά για τα οποία πολέμησαν οι προηγούμενες γενιές. Ε, τα παίζουμε όλα στον τζόγο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται να κρατήσουμε ζωντανέ τι ιδέε και τι αξίε πάνω στι οποίε στηρίζεται η Ευρώπη. και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το νέο αφήγημα δεν πρέπει να πετάξει το παλιό, αλλά πρέπει να το ξαναχρησιμοποιήσει. Να υπενθυμίσει δηλαδή στον κόσμο πού ε, χτίστηκε και πώς χτίστηκε η Ευρώπη, πού στηρίχθηκε. Πιστεύω λοιπόν πως η πιο σωστή μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσουμε τα υφιστάμενα, τα παλιά ε, συστήματα, τις παλιές δομές, να αλλάξει ίσως η δομή έτσι ώστε να γίνει πιο βιώσιμη, αλλά να ε, μην τα ξεχάσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάλινοφ θα ήθελα πραγματικά να σεβαστείτε το χρόνο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ε, σχεδόν ε, αγένεια θα ήταν να μην πάρω το λόγο σε αυτή τη συζήτηση, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να σας υπενθυμίσω ότι δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα διότι υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο ε, παρουσιάζουν οι αντιευρωπαϊστές ότι αγαπούμε την Ευρώπη, αγαπούμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά δεν μας αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ανυπεράσπιστοι ενώπιον αυτού του επιχειρήματος, αλλά θα ήθελα να τονίσω κάτι εδώ η μοναδικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μένα, ιδίω όταν ε, επικοινωνώ με νέους ανθρώπους που την ανταλαμβάνονται ως ευκαιρίες, ελευθερία και δικαιώματα. Και κατόπιν, βάσει αυτού του συμπλέγματος ευκαιριών, ελευθερίας και δικαιωμάτων, πηγαίνουν στις επιχειρήσεις, στην οικονομία, στον πολιτισμό. Και επομένως, πιστεύω, από την προσωπική μου πείρα, διότι έκανα κάτι αντίστοιχο για τρία χρόνια. Ο πιο εύκολος τρόπος ε, να πείσουμε τους νέους ανθρώπους είναι μέσω του διαλόγου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Διότι πολλοί από αυτούς δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον πολιτισμό, ίσως να έρθει αργότερα αυτό το ενδιαφέρον, αλλά αντιλαμβάνονται και θα έπρεπε να αντιλαμβάνονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μοναδικός χώρος ένα πολιτικό και νομικό επίτευγμα και ε, με αυτό ως υπόβαθρο μπορείς να απολαύσεις ε, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την πολιτισμική κληρονομιά, τις επιχειρήσεις και οτιδήποτε άλλο. Αυτά ήθελα να πω. Η κυρία Βόξερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτού που έλαβαν το λόγο προηγουμένω. Συμφωνώ ότι η επικοινωνία, ο διάλογο με του νέου ανθρώπου είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε του νέου ανθρώπου. Όταν δεν μιλούμε με του νέου ανθρώπου ε, και τι εμπειρίε του, ε, βλέπουμε ότι θέλουν οι ιδέε τους να υλοποιηθούν. Δεν θέλουν απλώς ε, όνειρα και φρούδε ελπίδες, θέλουν απτά αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω αυτό το πρόγραμμα για το νέο αφήγημα και σε συνέχεια των όσων ακούστηκαν να πω ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελεί δέλεαρ και προκειμένου να γίνει αυτό έχουμε δύο τρόπους. Ο ένας είναι η επικοινωνία, η βελτίωση της εικόνας της Ευρώπης αλλά δεν αρκεί να αναφερόμαστε στην εικόνα της Ευρώπης, πρέπει να τη βελτιώσουμε και πραγματικά την εικόνα. Πρέπει να κάνουμε πράξεις αυτά τα οποία πρεσβεύουμε. Πριν από 100 χρόνια η Ευρώπη ήταν η γη της επαγγελίας και επομένως αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να κάνουμε την Ευρώπη, να γίνει η γη της επαγγελίας, ε, η αμοιβαία αναγνώριση των ε, πτυχίων και των διπλωμάτων, οι πάρα πολύ σημαντικές ευκαιρίες να υπάρχει η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ούτω καθεξής. Εάν καταφέρουμε να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά, με πρακτικές ε, δράσεις και με μια βελτιωμένη εικόνα μπορούμε πραγματικά να έχουμε βελτιωμένες ε, προεπτικές. Ο κύριος Τζαμπάς και τελευταίος, ο οποίος θα είναι πολύ σύντομος με υποσχέθηκε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πράγματι πολύ σύντομος. Ήθελα να λάβω το λόγο διότι οι συνάδελφοί μου είπαν κάποια πράγματα αλλά εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στον ε, Επίτροπο δεν έχουν επιχειρήματα οι επιφυλακτικοί νέοι για τον ευρωσκεπτικισμό τους και αυτά τα επιχειρήματα έγκυνται στο γεγονός ότι και εμείς δημιουργούμε στερεότυπα. Ε, προωθούμε εθνικά ζητήματα Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, για παράδειγμα, δεξιοί, έχουν διαφορετικέ ιδεολογίε, αλλά είναι και Ευρωπαίοι. Δεν θα πρέπει να του καταδικάζουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι κατά τη Ευρώπη, γιατί το ευρωπαϊκό όραμα δεν είναι αριστερό, δεξιό, φιλελεύθερο ή συντηρητικό πρόγραμμα. Είναι ένα ευρωπαϊκό όραμα. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις αυτές και τώρα να δώσω το λόγο ε, σύντομα στον Επίτροπο. Να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ως όρος ο οποίος αναφέρθηκε σε πολλές από τις παρεμβάσεις σας, ο όρος γέφυρα. Ο πολιτισμός μπορεί να αποτελήσει το όχημα ε, που κατασκευάζει γέφυρες σε μια Ευρώπη που κατασκευάζει τείχη και υψώνει τείχη θα μπορούσε ως σύμβολο να είναι μια εικόνα που δίνει μια πολιτισμική προοπτική για αυτό το νέο αφήγημα και έτσι προσδίδεται μια πολύ σημαντική έννοια και είναι ουσιαστικό το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρώσουμε τη συζήτηση σε δύο επίπεδα. Μία μεταπολιτική συζήτηση, αν θέλετε, αυτό το νέο αφήγημα, το οποίο αναπτύσσεται βάσει ανοιχτή συζήτηση ε, σε χώρους ε, ε, και τρόπους που δημιουργούν μια νέα πολιτισμική διάσταση της φύσης της Ευρώπης, αλλά και που διασταυρώνονται και ενισχύουν όλες εκείνες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα προγράμματα τα οποία από την αρχική τους δομή θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα ευρωπαϊκή ηθαγένεια, μια νέα ευρωπαϊκή νοοτροπία και θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικές και πολιτιστικές πολιτικές θα πρέπει να προβάλλονται περισσότερο και θα πρέπει να δημιουργήσουμε και το κατάλληλο υπόβεθρο ώστε στη συνέχεια να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο θα ενισχύει αυτές τις διαστάσεις. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δούμε και με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε και καταρχάς να φροντίσουμε να εισακουστεί η φωνή μας αλλά και να συνεισφέρουμε σε αυτό το νέο στάδιο του αφηγήματος και οι γέφυρες φυσικά χτίζονται και μεταξύ γενεών. Και θα ήθελα και εγώ να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη από αυτού. Το είπε η συνάδελφο ε, Χιμένε Μπαρμπάτα αλλά και άλλοι συνάδελφοι. Δεν αφορά το θέμα μόνο του Ευρωπαίου πελίτε. Σήμερα πρέπει να αφηγηθούμε την Ευρώπη στον κόσμο. Εμεί αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμαστε ιδιαίτερα αξιόπιστοι ε, για κάποιε από τι ε, αξίε οι οποίε δεν είναι ιστερικέ αλλά είναι θεμελιώδει αξίε. Την αλληλεγγύη, την ελευθερία, τη δημοκρατία, τη συνεργασία στις στιγμές τις οποίες ε, ε, βιώνουμε. Στη Μεσόγειο, για παράδειγμα, δεν δείχνουμε ειλικρινά μία ταυτότητα και μία εικόνα τόσο συνεκτική, ε, πρέπει να ομολογήσω. Και νομίζω ότι αυτό το νέο αφήγημα, στο οποίο θα συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε αυτή την πολύ σημαντική ανακοίνηση που έκανε η υπατή εκπρόσωπος Μαγκερίνη με τον Επίτροπο Ναυράτσιτς και τον Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα γειτονίας, θα αποτελήσει και μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα νέο αφήγημα, αλλά και να προσδώσουμε ουσία στο όραμα της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο με τρίτες χώρες. Και αυτό θα είναι η μεγάλη πρόκληση, γιατί πλέον δεν απευθυνόμαστε μόνο στους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και σε όσους δεν γεννήθηκαν μεν στην Ευρώπη, αλλά ζουν στην Ήπειρο και θέλουν και αυτοί να χτίσουν γέφυρες προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Το κάναμε και με την κατεστραμμένη πολιτισμική κληρονομιά, αλλά θα πρέπει να χτίσουμε και άλλες γέφυρες οι οποίες ε, γκρεμίστηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ναβράτσιτς, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς όλους για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Ε, θα μας είναι πολύ χρήσιμα για τη μελλοντική μας δουλειά καθώς θα αναπτύσσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις για το νέο αφήγημα. Έχω απόλυτη επίγνωση των ζητημάτων που υπάρχουν στον ορίζοντα 2020 και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και κάνουμε αυτή τη στιγμή ό,τι μπορούμε και με τους ε, άλλους επιτρόπους για να ε, τα διορθώσουμε. Γνωρίζω πως ε, υπάρχει στήριξη ε, παρόλες τις δυσκολίες για το ορίζοντας 2020 και για τους ε, εκπαιδευτικούς από την ε, και από την Ανατολική Ευρώπη. Προσπαθούμε μέσω του ΕΦΣΥ να βοηθήσουμε το θέματα της εκπαίδευσης. Και θα ήθελα τώρα να ε, επικεντρωθώ στα βασικά σημεία αυτού του νέου αφηγήματος. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι η τελευταία ηλικιακή ομάδα που έχω πρόθεση να ξεχάσω είναι η ηλικιωμένη, γιατί και εγώ προς τα εκεί οδεύω. Ναι, αν πρέπει να διαλέξουμε ένα μόνο μικρό κομμάτι όλου του ε, οικοδομήματος της Ευρώπης, αναπόφευκτα θα θέσουμε προτεραιότητες. Γι' αυτό λοιπόν θα επισκιαστούν ορισμένα άλλα θέματα. Συμφωνώ όμως απόλυτα μαζί σας για το ότι δεν υπάρχει μέλλον χωρίς ε, αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, χωρίς γέφυρες ανάμεσα στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Αλλά, αν δούμε τις πολιτικές εξελίξεις μόνο από αυτή τη βδομάδα, από τις τοπικές εκλογές στην Ιταλία, από τις πρόορες εκλογές στην Κροατία, στην Ισπανία και φυσικά ε, με το Βρετανικό δημοψήφισμα, θα δούμε ότι αυτά είναι σημάδια δυσπιστίας. Σημάδια δυσπιστίας προς τους πολιτικούς. Πως ε, υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στην πολιτική ελίτ και στους πολίτες Δυστυχώς όμως υπάρχουν και βαθύτερα χάσματα, ρήγματα θα έλεγα, ανάμεσα στου ίδιου του πολίτε. Και αυτό πιστεύω πως είναι το πρόβλημα. Ο κατακαιρματισμό της ε, σημερινής ευρωπαϊκής κοινωνίας, ο ατομισμός που υπάρχει και στους πολίτες και στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό χρειάζεται οι κοινότητε και οι κοινωνίε να είναι ενωμένε, να είναι ισχυρέ και να χτίσουμε το μέλλον μα πάνω σε αυτέ. οι νέοι είναι μία κοινότητα από μόνοι τους. Είναι μία αφηρημένη έννοια διότι είναι κατακαιρματισμένη ανάλογα την περιφέρεια, τη χώρα, την περιοχή, την πόλη κτλ. Όμως, λόγω της ε, διαφορετικότητας που υπάρχει στις τεχνικές επικοινωνίας, στις γλώσσες, στην ε, γεωγραφική κατανομή, υπάρχει ένας κοινό παρανομαστής. Όλοι δηλαδή έχουν κοινά σημεία αναφοράς, κοινούς ε, ήρωες, κοινά ενδάλματα. Αν λοιπόν εστιάσουμε σε αυτούς και προσπαθήσουμε να τους καταλάβουμε, ίσως βρούμε μία λύση για την Ευρώπη. Δεν θα έλεγα ότι το νέο αφήγημα είναι μία πρόταση και ότι είναι η πρόταση που θα έχει αποτελέσματα. Είναι μία δυνατότητα. Φυσικά και δεν είμαι αισιόδοξο για το ότι θα βρούμε μία λύση που θα ταιριάζει σε όλε τι περιπτώσει, διότι αλλάζουν τα πάντα με ταχύτητα του ρυθμού. Όμω το νέο αφήγημα μα παρέχει μία πλατφόρμα για συζήτηση. Μια πλατφόρμα για τη νεολαία. Και αυτό πιστεύω είναι το πρώτο στάδιο. Πρώτα χρειάζεται δηλαδή να βρούμε μια κοινή γλώσσα να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο. Ένα κοινό πλαίσιο κατανόησης για το τι γίνεται σήμερα στην Ευρώπη. Γιατί εδώ πιστεύω πως υπάρχει διαφωνία. Εδώ πιστεύω πως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για την σημερινή κατάσταση της Ένωσης, για το ποιες είναι οι αιτίες της κρίσης, για το αν η κρίση είναι οικονομική, πολιτική, κοινωνική ή κρίση αξιών, η κριση αξιων ταυτότητας. Εάν λοιπόν γίνει μία ευρύτατη ανταλλαγή απόψεων, μία μεγάλη διαβούλευση και εντοπίσουμε τα σημεία στα οποία υπάρχει συνένεση και τα σημεία στα οποία υπάρχουν αποκλήσεις, αυτό πιστεύω είναι εξίσου ε, σημαντικό, ε, παρεμπιπτόντως, οι διαφωνίες με τις συμφωνίες, τότε θα έχουμε βρει έναν κοινό τόπο για να χτίσουμε ένα κοινό μέλλον. Και αυτό είναι ο ρόλος του νέου αφηγήματο. Να συλλέξει δηλαδή τις ε, απόψεις των εκπροσώπων της νεολαίας και μετά να καταλάβουμε τα προβλήματά τους. Είναι μία γενιά με πολλές δυσκολίες, είναι μία γενιά που μαστίζεται από ανεργία. Μία γενιά όμως που είναι ε, αφιερωμένη στην Ευρώπη, δεσμεύεται και την Ευρώπη. Αν δείτε ανάμεσα στους νέους ποιες είναι οι πολιτικές ε, πεπιθήσεις, θα δείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα ότι οι νέοι είναι πιο κοντά στην Ευρώπη από ότι οι άλλες ομάδες. Είναι λοιπόν μια τεράστια ευκαιρία να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πρώτα όμως πρέπει να καταγράψουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν, τους κινδύνους. Γι' αυτό λοιπόν ε, εδώ θα σταματήσω και θα σας πω κλείνοντας ότι σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας, όλους όλα τα μέλη και τους πρέσβεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ όλους τους πρέσβεις για τη συνεισφορά σας, ευχαριστώ πολύ και όλους τους συναδέλφους. Φαντάζομαι πως θα πρέπει και να συμφωνήσουμε, να υπάρξει μια συμμαχία για ένα κοινό ευρωπαϊκό κανάλι. Διότι όπως είπατε, είναι πολύ σημαντική η, ε, ναι, είναι πολύ σημαντικά τα προγράμματα για αυτούς. Πρόσφατα συναντήθηκα με ε, τον ε, πολιτισμικό διευθυντή ενός μεγάλου Καναλιού στην Ιταλία και αυτά άκουσα. Τα ίδια που λέμε και εδώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ όλους και ας συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη μετά από ένα λεπτό διάλειμμα για να αποχαιρετήσω τους προσκεκλημένους μας.

Υπότιτλοι Λοιπόν, ε, τώρα έχουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία την οποία προωθήσαμε και θέλουμε να αφιερώσουμε αυτό το τελευταίο τμήμα της συνεδρίασής μας στον αθλητισμό. Θεωρώ ότι υπάρχει ε, μεγάλη ανάγκη να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό, να ξεκινήσουμε και μια πολιτική πρωτοβουλία για τον αθλητισμό και να εμβαθύνουμε στα διάφορα θέματα ε, για τα οποία θα πρέπει να κάνουμε και πιο προηγμένες προτάσεις. Γνωρίζουμε... σημαίνει κάτι? Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι ε, θα γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, καταρχάς ε, για τον τομέα του αθλητισμού στα πλαίσια της έκθεσης που έχει αναλάβει ο συνάδελφος Τάκουλα για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ε, πολιτική για τον αθλητισμό και έχουμε θέσει ως θέματα την καλή διακυβέρνηση για την προσβασιμότητα και την ακαιρεότητα με τη συμμετοχή και κάποιων άλλων εισηγητών. Ε, με αυτή την ανταλλαγή απόψεων ε, ξεκινάμε και τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τον Αθλητισμό που θα γίνει το Σεπτέμβριο, αλλά θα είναι την εβδομάδα που θα είμαστε στο Στρασβούργο. Ε, σας προσκαλώ και σε μια έκθεση που θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα περί τίνος πρόκειται, αλλά δεν είναι ακριβώ έργο της Επιτροπής. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Εύα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το να μιλάμε για κεραιότητα του αθλητισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό δεδομένων και των όσων συμβαίνουν. Θα είδατε και για τον αποκλεισμό της ε, ρωσικής ομάδας από τους Ολυμπιακούς για λόγους ε, ντόπινγκ ε, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα το οποίο ε, φαίνεται να είναι ε, υπό τη δικαιοδοσία των διεθνών συμβάσεων. Χρειάζεται όμως ε, και περαιτέρω δράση από πλευράς μας, όπως επίσης και το θέμα της πρόσβασης και του διεθνούς αθλητισμού, που είναι ένα άλλο ζήτημα. Έχουμε λοιπόν αυτό το πάνελ ομιλητών και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους εμπειρογνώμονές μας και μετά από την εισαγωγή του κυρίου Τάκουλα θα τους δώσουμε φυσικά το λόγο και ε, θα δώσουμε φυσικά και στους κοιόδης συζητητές. Έχουμε τον κύριο Αλεξάνδερ Χάστινγκ, ο οποίος είναι πρώην επικεφαλής της ομάδας ε, του Συμβουλίου για τον Αθλητισμό, ε, πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας του Αθλητισμού, τον Τάπιο Κόρους, ο οποίος ήταν ε, ε, πρωταθλητής στο Ακόντιο ε, Φιλανδός και τον κύριο Ιβλε Λοστέκ από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος ε, ανέκαθεν ήταν από τους θαμώνες εδώ στην Επιτροπή μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την παρέμβαση του συναδέλφου Τάκουλα για να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση και μετά θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα σας τα πω στα φιλανδικά, που είναι και η μητρική μου γλώσσα. Έντεκα χρόνια μέλος στην Επιτροπή Πολιτισμού έχω δει πολλά και ποικίλα πράγματα και βεβαίως και σχέση με τον αθλητισμό, ιδίως με τη Λευκή Βίβλο σχετική με τον αθλητισμό και θεωρώ ότι είναι προνόμιο που ε, μου ανατίθεται το θέμα του αθλητισμού σε αυτό το σημαντικό έτος για τον αθλητισμό. Έχουμε φέτος διάφορες σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις, το, Ευρωπαίο, ε, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, τους ε, αγώνες στην Βραζιλία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και ο αθλητισμός βεβαίως είναι γνωστό ότι έχει και σημαντικές θετικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Η έλλειψη αθλητικής δραστηριότητα ε, οδηγεί σε πρόωρους θανάτους. Χρειάζεται λοιπόν πολιτική για τον αθλητισμό. Εγώ έρχομαι σε τέσσερα βασικά θέματα. Στον αθλητισμό πρώτα την ακαιρεότητα, προσβασιμότητα και όλα τα σχετικά θέματα. Ως αφετηρία ε, λαμβάνω μια πυραμιδωτή διάρθρωση του αθλητισμού. Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί η πολιτική του αθλητισμού. Έχουμε δει ποικίλα σκάνδαλα στα αθλητικά, τα οποία δίνουν κακό παράδειγμα και υπονομεύουν την ε, καλή φήμη του αθλητισμού. Χρειαζόμαστε διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων. Χρειαζόμαστε ε, επίσης διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις πηγές χρηματοδότησης. Χρειάζονται ξεκάθαρα κριτήρια και αυτά να εφαρμόζονται σε όλες τις πηγές χρηματοδοτήσεως. Πάλι εδώ το, ε, ο αθλητισμός στην βάση είναι πάρα πολύ σημαντικός. Στην έκθεσή μας εξετάζουμε σχετικά θέματα, ε, σχετικά με την ακαιρεότητα, σχετικά με βία γεγονότα ε, που σημειώνονται στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και ζητούμε μηδενική ανοχή απέναντι σε εκδηλώσεις ρατσισμού, βίας και φασισμού. Έχουμε ακούσει βέβαια και τα σχετικά με το ντόπινγκ και εκεί πρέπει να φανούμε πολύ σκληροί και απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια χειραγώγησης. Σημαντικό και αυτό λοιπόν στην πολιτική αθλητισμού. Χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να συμμετέχει στα αθλητικά και βεβαίως να φροντίσουμε και για ανθρώπους που έχουν ειδικέ ανάγκες και τη δυνατότητά τους να ασκήσουν αθλήματα. Και αυτά πρέπει να περιληφθούν και βεβαίως να μπουν και στα σχολεία. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση προσφύγων, μεταναστών, για την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στις κοινωνίες. Πρέπει να στηρίξουμε τον αθλητισμό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίως να στηρίξουμε αυτούς που επιθυμούν να κάνουν σταδιοδρομία στον αθλητισμό το Erasmus Συν, το Erasmus Plus, παίζει σημαντικό ρόλο εν προκειμένου και μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντικό εφαρτήριο, ιδίως για τους ε, προπονητέ. Θα επανέλθουμε σε αυτά. Οι συνάδελφοί μου καλούνται να συμβάλλουν και αυτοί με τις ε, τροπολογίες τους και τα άλλα σχετικά στην προσπάθεια εκπόνησης εκθέσεως. Πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Αλεξάνδρ Χάστινγκ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριο Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση να σας ε, παρουσιάσω τις απόψεις μου για τον αθλητισμό, για την ε, έκθεσή σας, για την πολιτική αθλητισμού. 5 με 10 λεπτά είναι πρόκληση για μένα. Νιώθω σαν την Πινελόπη του Οδυσσέα ε, που ε, θα ε, ξυλώσω, μάλλον θα, θα φτιάξω σήμερα, θα εφάνω σήμερα αυτό το οποίο ξετήλησε χθε το βράδυ. Πρέπει να αναφερθούμε στην καλή διακυβέρνηση και στην προσβασιμότητα. Θα μιλήσω στα γαλλικά, παρά το γεγονός ότι η παρουσίασή μου είναι στα αγγλικά, γιατί θα με διευκολύνει. Δεν είχα και πολλές δυσκολίες για να ετοιμάσω την παρουσίασή μου για σήμερα, διότι το μόνο που είχα να κάνω είναι να παρακολουθώ τηλεόραση τους τελευταίους μήνες. Ε, περιστατικά διαφθοράς ε, για υφήνοντες ε, διεθνών οργανώσεων. Η διαφθορά ήταν και μια ιδιαίτερη μέθοδος διακυβέρνησης. Υπήρχαν επίσης περιστατικά ντόπινγκ που περιελάμβαναν και διαφθορά, χειραγώγηση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων και αναφέρθηκε ήδη και ε, κάποια περιστατικά βίας ε, τα οποία ασκούν ε, συγγνώμη, βία η οποία ε, προέρχεται από φιλάθλους σε πρόσφατες αθλητικές εκδηλώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ενισχυμένη συνεργασία προκειμένου να βελτιώσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δημοσίων αρχών και αθλητικών ιδιωτικών αρχών και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα διάφορα ε, δίκαια ε, συμβάσεις ε, που αφορούν τη διαφθορά, το στήσιμο των αγώνων και το ντόπινγκ. Ε, θα πρέπει επίσης ε, να δούμε και τι γίνεται με τις υποψίες διαφθοράς ε, για τις διάφορες διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και θέματα προς σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ευρωπαϊκών αξιών κατά την διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, πράγματα τα οποία βρίσκονται στην επικυρότητα, δικαιώματα των εργαζομένων, ανηλίκων, γυναικών, ομοφιλοφίλων κ.ο.κ. Στη συνέχεια. Όσον αφορά την προσβασιμότητα. Ε, και εδώ δεν δυσκολεύτηκα ε, βλέποντας τι γίνεται στην τηλεόραση και παρακολουθώντας ένα διεθνή ποδοσφαιρικό αγώνα ε, με κάποιους οι οποίοι πριν από 20 χρόνια θεωρούνταν πρόσφυγες ενώ τώρα είναι οι διεθνείς παίκτες της Αυστρίας, της Σουηδίας ή της Κροατίας. Αυτό καταδεικνύει ότι αφενός ο αθλητισμός και η αυτή ζέση που μπορεί να προκαλέσει σε αυτούς τους ε, πρώην πρόσφυγες μπορεί να αλλάξει την εικόνα που μπορεί να έχουν οι Ευρωπαίοι ενώπιον των προσφύγων και αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός είναι ε, συντελεστής ε, ένταξης και κοινωνικής αφομοίωσης. Πέραν των όσων διαπίστωσα πρόσθεσα, ε, πρόσφατα παρακολουθώντα ε, την τηλεόραση, υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να αναφέρουμε όσον αφορά την ακαιρεότητα. Υπάρχει το ευρωπαϊκό μοντέλο του αθλητισμού, το οποίο αμφισβητείται ιδιαίτερα σε διάφορα επίπεδα από την ε, Διεθνή Οργάνωση του Πατινά και από τη Διεθνή Οργάνωση Καλαθόσφαιρα, αλλά δεν θα επισέλθω σε περισσότερε λεπτομέρειε. Υπάρχει υπόθεση ESU στα πατινά ταχύτητα και τον υπάρχουν κλειστά γήπεδα μπάσκετ. Ε, προωθούμε την εξαφάνιση της αρχής της προώθησης, αλλά προσπαθούμε επίσης ε, να έχουμε ένα σύστημα οικονομικής αλληλεγγύης μεταξύ των βασικών αθλημάτων, των ερασιτεχνικών αθλημάτων και των επαγγελματικών αθλημάτων. Υπάρχουν επίσης ε, κάποια στοιχεία για τα όσα αναφέρομαι την, ε, τρίτη ιδιοκτησία που απειλούν και τον ανταγωνισμό αλλά και τον, ε, ε, την προσωπική αξιοπρέπεια των αθλητών. Υπάρχει η αύξηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό που είναι ένας από τους καλούς λόγους να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού που θα προωθήσει και τη φυσική δραστηριότητα αλλά και τον εθελοντισμό στον αθλητισμό. Ε, η σύνθεση των εθνικών ομάδων είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε επίση και στα θέματα τη χρηστή διακυβέρνηση υπάρχει και το γεγονό ότι υπάρχουν ολοένα και περισσότερε απαιτήσει από του αθλητικού ομίλου για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Ολοένα και μεγαλύτερα στάδια, ε, πολύ περισσότερε τεχνικέ απαιτήσει και οικονομικά μοντέλα διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων που τελικά, εάν προσέξουμε, βλέπουμε ότι τα ουσιώδη δεν ε, τα περιλαμβάνουν, ενώ το κόστος ε, το αναλαμβάνει ουσιαστικά το δημόσιο. Όσον αφορά την ε, προσβασιμότητα, και με αυτό θα ολοκληρώσω, όσον αφορά στη χρηματοδότηση, νομίζω ότι σε θέματα χρηματοδότησης η οργανώσεις καταπολέμησης του ντόπινγκ και κατά της της διαφθοράς ε, μας δείχνουν ότι πρέπει να έχουμε νέους τρόπους χρηματοδότησης του αθλητισμού ε, και χρειαζόμαστε και τρόπους χρηματοδότησης που πρέπει αφενός ε, να βοηθήσουν και τους χορηγούς και τους διεθνείς ομοσπονδίες αθλητισμού και το καθεξής. Πέρα λοιπόν τη χρηστή διακυβέρνηση και τη ακαιρεότητα, μα ενδιαφέρει και η οικονομική ε, ανεξαρτησία των ε, αθλητικών εκδηλώσεων. Φαίνεται ότι αυτό που έχει τα περισσότερα χρήματα τελικά κερδίζει και το πρωτάθλημα. Ε, όσον αφορά την προσβασιμότητα και τα σχετικά θέματα, έχω διακρίνει δύο κατηγορίες προσβασιμότητας. Η μία είναι η προσβασιμότητα των ατόμων, στον αθλητισμό και στην ε, διοργάνωση και διαχείριση του αθλητισμού. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που περιλαμβάνει τις γυναίκες, ε, τους ε, ΛΟΑΔ, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, φυλακισμένους, ε, Πρόσφυγε και μετανάστες. Ε, δεν θα επιστρέψω σε λεπτομέρειε. αλλά φαίνεται ότι οι κοπέλες ε, κάνουν λιγότερο αθλητισμό και συμμετέχουν λιγότερο σε αθλητικές εκδηλώσει. Είναι πολύ δύσκολο να εντάξουμε ένα πρόσφυγα σε επίσημη εκδήλωση αν δεν έχει επίσημη άδεια από τον αρχικό του σύλλογο και είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ένα σύστημα διπλής καριέρας για κάποιον ο οποίος δεν είναι υπήκος μιας χώρας. Υπάρχει και το θέμα της ε, προσβασιμότητας των ανηλίκων. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο και πολύ σημαντικό. Αφορά και την προστασία κατά της ε, φυσικής κακοποίησης, ε, της σωματικής κακοποίησης, και το να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και επίσης και το πάρα πολύ σημαντικό θέμα του αθλητισμού των νέων και των πολύ μικρών παιδιών από το παιδικό σταθμό, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Όσον αφορά τα θέματα αυτά της προσβασιμότητας, θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται ε, με το τι κάνει ο αθλητής μετά την επαγγελματική του σταδιοδρομία, αν υπάρχουν μηχανισμοί να αλλάξει επάγγελμα και επίσης κατά την άποψή μου θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα της ε, πρόσβασης στον επαγγελματικό αθλητισμό που αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία ρύθμιση, δεν το συζητούμε πια αλλά υπάρχουν ε, προβλήματα. Άλλο ένα θέμα όσον αφορά την προσβασιμότητα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε είναι η αναγνώριση στην Ευρώπη επαγγελματικών προσόντων, πιστοποιητών. Ε, πτυχίων κλπ. Ε, εκπαιδευτών, προπονητών και ούτω καθεξής. Ε, και επίσης έχουμε, όπως σας είπα, την προσβασιμότητα των ατόμων. Δεν ξέρω αν είναι τόσο σημαντικό αυτό για την έκθεσή σας, αλλά μπορεί να υπάρχει και προσβασιμότητα σε αθλητικές εκδηλώσεις. Εδώ υπάρχουν θέματα δικαιωμάτων, αναμετάδοσης, πρόσβαση σε περιεχόμενο και ούτω καθεξής και χωρίς να θέλω να επηρεάσω την έκθεσή σας ή τον τρόπο με τον οποίο θα συνταχθεί, αλλά θεωρώ ότι σε αυτή την έκθεση θα ήταν σημαντικό να ε, πάμε στην καρδιά των θεμάτων που δεν έχουν αναλυθεί ακόμα. Όσον αφορά το θέμα του αθλητισμού, υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση των βασικών προβλημάτων. Γνωρίζουμε όλοι τον ντόπινγκ, τη διαφορά, το στήσιμο αγώνων, αλλά υπάρχουν και κάποια θέματα επί των οποίων θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Για παράδειγμα, η διπλή ε, καριέρα ε, ένας φοιτητής που τώρα θέλει να πάει στο εξωτερικό για να ασκείται και να αθλείται, ε, είναι σχεδόν αδύνατο να το επιτύχει ε, εάν δεν ανήκει σε κάποιον ε, αθλητικό όμιλο του εξωτερικού και αυτό είναι δύσκολο γιατί θα είναι ανταγωνιστής ε, σε σχέση με την προηγούμενη του ομάδα. Ε, όσον αφορά τη βία, έχουμε διαπιστώσει όλοι περιστατικά βίας και θα έπρεπε ίσως να υπάρχει ένα διεθνές μητρό που να καταγράφει αυτά τα γεγονότα. Και τέλος θεωρώ ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται, κατά την άποψή μου, στα πλαίσια των συγκεκριμένων ε, ορίων σε συνεργασία με τον κόσμο του αθλητισμού και βάσει και των ορίων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι μπορεί να κάνει. Και όσον αφορά τον αθλητικό κόσμο, ε, τον επικρίνουμε ε, ναι μεν και δικαίως ορισμένες φορές, αλλά δεν είναι ο μόνος ο οποίος υπερασπίζεται τον αθλητισμό με αξίες, με αλληλεγγύη, με ευγενή άμυλα ε, και δεν υπάρχουν μόνο εμπορικά συμφέροντα τα οποία πολλούνται και αγοράζονται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χάστινγκ για αυτή την πολύ ωραία παρουσίαση η οποία ε, συνοπτικά μας έδωσε κάποια στοιχεία ε, με απόλυτη ειλικρίνεια. Ανηλέησε ορισμένε φορές αλλά ήταν πολύ σημαντικά όλα αυτά αμέσως μετά, γιατί σας είπα ότι το απόγευμα αυτό το έχουμε αφιερώσει στον αθλητισμό, θα έχουμε την ε, παρουσίαση μιας έρευνας που ζητήσαμε από το Τμήμα Μελετών για ε, τη δυτή καριέρα στον αθλητισμό. Θα σας τη δώσουμε αμέσως. Υπάρχουν αντίγραφα για να δείτε ότι αυτά τα οποία αναφέρετε εσείς ως ε, θέματα πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος για τους νέους αθλητές πραγματικά είναι θέματα που μας απασχολούν και εμάς και έχουμε εμβαθύνει από αυτό. Να δώσουμε τώρα το λίγο στον κύριο Τάπιο Κόριους, ε, πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Ομάδας Αθλητισμού. Παρακαλώ. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta saapua tähän kuulemista. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Ο αθλητισμός είναι ένας χώρος ο οποίος επεκτείνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο. Και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε ορισμένα ζητήματα και να δώσουμε απαντήσεις. Πώς θα πρέπει να είναι η πολιτική για τον αθλητισμό μπορώ να σκεφτώ ε, τα εξή. Καταρχάς, ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Είναι κάτι που κάνεις εφόρου ζωής. Είναι ένας τρόπος ε, για να έχεις υγεία, για να έχεις ευεξία. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε ότι δεν αθλούμαστε αρκετά, ότι κάνουμε καθιστική ζωή. Έπειτα, είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τα χαρίσματα που έχουν οι νέοι άνθρωποι. Να στηρίξουμε λοιπόν τον αθλητισμό και τους επαγγελματίες αθλητές έτσι ώστε να εξελιχθούν. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το διπλό σύστημα για μένα είναι πάρα πολύ χρήσιμο ο αθλητισμός είναι και επαγγελματική στα διαδρομία, αρκετά σημαντική. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις πτυχές ε, του αθλητισμού όταν προσπαθούμε να χαράξουμε πολιτική για τον αθλητισμό, να δούμε οριζόντια το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε συνεργασίες, αλλά και σε κάθε το επίπεδο πολιτικής να δούμε πώς οι διεθνείς οργανισμοί θα διέπονται από, ίδιους, από τους ίδιους κανόνες και από τις ίδιες αρχές. Χρειάζεται επίσης να βρεθούν κανόνες οι οποίοι θα ισχύουν σε όλο τον κόσμο και θα διασφαλίζουν καθαρό αθλητισμό Ας μην ξεχνάμε όμως ότι και ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ κοντά στον άνθρωπο που μπορεί να γίνει και, ε, και στο σπίτι μας. Ε, μπορεί να γίνει στο σπίτι μας με την οικογένειά μας, σε κάποιον αθλητικό σύλλογο, έξω στη φύση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι δηλαδή για να αθληθεί κανείς. Θα έλεγα ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε την ε, συζήτηση σε όλο τον κόσμο για το πώς μπορούμε να αλληλοβοηθηθούμε, πόσο οι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί θα ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, αλλά και θα δημιουργήσουν κοινούς κανόνες για τον αθλητισμό. Φυσικά, πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλοι κλάδοι, όπως η εκπαίδευση. Πρέπει να μιλήσουμε για το περιβάλλον, για τον πολιτισμό, για την νεολαία. Και πρέπει να γίνει λοιπόν αυτή η πολυεπίπεδη συζήτηση και σε επίπεδο τοπικής ε, περιφερειακής αυτοδιοίκησης για να αποκομίσουμε μία ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει και του τι πρέπει να γίνει στο μέλλον με τον αθλητισμό. Κάτι άλλο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι οι πόροι, η χρηματοδότηση. Και θα ήθελα να κοιτάξουμε τριών ειδών πόρους, ε, τι, τους πόρους τους οποίους μπορούμε εμείς να συνεισφέρουμε. Και λοιπόν, χρειάζεται να συμπεριληφθούν όλοι, χωρίς αποκλεισμούς. Ο καθένας μας μπορεί να λάβει αποφάσεις για τον εαυτό του, μπορεί να αποφασίσει πόσο θα ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Μπορεί ο νέος να αποφασίσει πώς θα ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Ο ηλικιωμένο επίσης, όλα τα μέλη της κοινωνίας. Επίσης, χρηστή διοίκηση είναι κάτι εξίσου σημαντικό. Χρειάζεται χρηστή διοίκηση, η σωστή ηγεσία και ο συνάδελφος πριν ανέφερε κάποια παραδείγματα για το αντίθετο κακοδιοίκησης όπως με τα πρόσφατα γεγονότα. Επίσης, εκπαίδευση. Η εκπαίδευση παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και χρειάζεται λοιπόν να της δώσουμε τη δέουσα προσοχή. Αυτό ήταν ο πρώτος κλάδος, το πρώτο σύνολο. Δεύτερον, οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα ε, διεξάγονται οι αθλητικές οργανώσεις, οι προϋποθέσεις από τις οποίες θα αθλούμαστε. Υπάρχουν διάφορες διασυνδέσεις με τις τοπικές αρχές, με τους συλλόγους, υπάρχουν ιδιαιτερότητες από χώρα σε χώρα και πρέπει να δώσουμε τη δόση προσοχή. Για παράδειγμα, διάφορα αθλητικά κέντρα, παιδικές χαρές. Είναι εύκολο για τα παιδιά να βγουν έξω και να αθληθούν, να το κάνουν δωρεάν. Εάν είναι δωρεάν, εάν υπάρχει κοντά κάποιο αθλητικό κέντρο, κάποιο πάρκο για skateboard, για parkour, τότε μπορούν να έρθουν πιο κοντά στον αθλητισμό οι νέοι. Έπειτα, χρηματοδότηση. Χρειάζεται χρηματοδότηση και από δημόσιους φορείς και από ιδιωτικούς. Και εδώ φυσικά πρέπει να μιλήσουμε και για την νομοθεσία, για τη φορολογία, για την νομοθεσία που θα διέπει την υγεία, το περιβάλλον, όλα αυτά τα θέματα που άπτονται του αθλητισμού. Αυτό φυσικά συνεπάγεται και διεθνείς κανόνες για τον αθλητισμό και χρειάζεται συμφωνία. Χρειάζεται να βρεθεί το πώς θα βελτιωθεί η χρηματοδότηση και να, βρεθούν πολλές πηγές χρηματοδότησης. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσω και να αναφερθώ σε κάτι το οποίο δεν ε, αναφέρεται συχνά τους θεατές. Τους θεατές ε, σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις, τους ε, συμμετέχοντες επίσης, τα συμμετοχικά αθλήματα, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι ανεξάρτητα από την ηλικία τους, να διασκεδάσουν και να βελτιώσουν την υγεία τους. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χρηστή διοίκηση, να υπάρχει σωστή ηγεσία και ο αθλητισμός να είναι κάτι το οποίο θα αφορά όλους και ας μην ξεχνάμε τους πολίτες, τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων ε, των προσπαθειών μας. Σας ευχαριστώ. εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά μας παίζει και λίγο χρόνος. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όμως η παρέμβασή σας. Και εγώ άλλωστε θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε δύο διαφορετικούς στόχους, ε, τις μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις και τα αθλήματα που έχουν κυρίως ε, θεατές και φιλάθλους και ε, ο αθλητισμός ο οποίος ε, ε, προλαμβάνει τη βία και την ευγενή άμυλα και όχι την επιθετικότητα. Αναφερόμαστε λοιπόν στην αθλητική δραστηριότητα ως μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λελοστέκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά. Και πρώτα επιθυμώ να πω ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε ε, πολύ ευνοϊκά την ιδέα της εκθέσεως για τον αθλητισμό, την ακαιρεότητα, την ε, ισότητα και την καλή χρηστή διοίκηση ή διαχείριση. Είχαμε και παλαιότερα την εκθεσή φύσας που είχε πολύ βοηθήσει και είχε εμπνεύσει πολλές δράσεις οι οποίες ανελήφθησαν εκ των υστέρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ αυτών και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των ε, Αθλημάτων στην οποία είχε συμμετάσχει ενεργά και ο προλαλή σας. Προσεγγίζουμε με πολύ φιλόδοξο τρόπο την έκθεση. Άλλωστε ο χρονισμός της εκθέσεως είναι εξαιρετικός. Ο εισηγητής έχει και μεγάλη τύχη διότι η έκθεσή του αυτή λόγω του χρόνου που έχει επιλέξει έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει. Αν κατανοώ καλά θα εγκριθεί επισήμως ίσως ε, στις αρχές του επόμενου έτους. Άρα σε μια περίοδο που θα συζητείται το, ο σχεδιασμός της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2020 για το πρόγραμμα Erasmus ε, Plus, ειδικό στον αθλητισμό, άρα θα έχει μεγάλο δυναμικό επηρεασμό και θα τροφοδοτήσει και τις εκθέσεις που θα έρθουν από τις δύο ομάδες υψηλού επίπεδου μετά από πρωτοβουλία του Επιτρόπου Ναύρατσιτς, την, ε, την αθλητική διπλωματία δηλαδή, <clears throat> μεταξύ αυτών. Τα λέω όλα αυτά για να εξηγήσω ότι πράγματι το timing είναι εξαιρετικό θα επιτρέψει στην έκθεση να έχει πολύ μεγάλη επιρροή. Πολύ σύντομα τώρα το αντικείμενο ή τα αντικείμενα που θίγει η έκθεση, ο, Επίτρο, ο εισηγητής κ. Στάκουλα ε, αναφέρθηκε στα πιο σημαντικά ζητήματα, δηλαδή πρώτα-πρώτα της ε, διοίκησης ή διαχείρισης. Governance. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να συμβάλλουμε μέσα στα πλαίσια που εξήγησε ο ε, συναδελφός μου Αλεξάνδρου Στίνγκ να συμβάλλουμε λοιπόν και στη διοργάνωση των ε, αθλητικών εκδηλώσεων κλπ. Και βεβαίως στις 15 Σεπτεμβρίου ο Επίτροπος Ναύρατσιτς θα συγκαλέσει διάσκεψη για την σωστή διαχείριση των αθλητικών. Θίξατε και το ζήτημα της διπλής σταδιοδρομίας την συμφιλίωση των εισαγωγικών του αθλητισμού και της επαγγελματική σταδιοδρομίας ή αθλητισμού και σπουδών. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πολύ. Θυμούμε η υπολουξεμβουργική προεδρία ένα συνέδριο όπου ένας αθλητής ε, Λουξεμβούργιος είχε πει εγώ σπουδάζω στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχω όμως την ίδια πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις όπως οι Βρετανοί που συναγωνίζονται μαζί μου. Το ίδιο συμβαίνει, μου είπαν αυτοί, και για όσου σπουδάζουν, για παράδειγμα, στη Γαλλία και αλλού. Επομένω, πρόσβαση, η προσβασιμότητα, η κινητικότητα επίση είναι σημαντικό, διότι στο έρασμό συν αθλητισμό δεν υπάρχει κινητικότητα. Είχαμε επιλέξει την προσέγγιση αυτή παλαιότερα, διότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα. Όμω θα συνταχθεί έκθεση η οποία θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε την ιδέα που νομίζω ότι είναι και κλειδί για την προώθηση της ε, ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού. Για κεραιότητα, Ο συνάδελφος μου Αλεξάνδρ αναφέρθηκε σε μια σημαντική διάσταση. Υπάρχει η Διεθνή Σύμβαση του ε, Συμβουλίου της Ευρώπης για το match fixing και για το doping. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται με διαφόρους τρόπους στις συζητήσεις αυτές. Υπάρχει, όπως είπα, η σύμβαση που έχει μάλιστα κυρωθεί για το μαγείρεμα των αγωγικών των αθλητικών αγώνων και τέλος για την προώθηση του αθλητισμού βάσεως και εκεί έχουμε φιλόδοξα σχέδια. Το έρασμο ΣΥΝ προβλέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον αθλητισμό βάσεως. Χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα πράγματα και αναμένουμε τις ιδέες που θα προβληθούν και από την έκθεση σας αυτή για να δούμε πώς θα προωθήσουμε τον αθλητισμό βάσος. Θα αρκεστώ σε αυτά. Θεωρώ ότι μπορώ να αρκεστώ στην, για την ώρα να ε, αναφερθώ δηλαδή στην διάθεσή μας να συμβάλλουμε στην σύνταξη της εκθέσεως. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λελοστέκ. Εμείς συμφωνούμε απολύτως ότι πράγματι έχουμε πλέον μια πολύ σημαντική βάση που αποτέλεσε και το έναυσμα για πολιτικές από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρχε η έκθεση ΦΥΣΑΣ ε, στην οποία ε, συνεισέφερε όλη η Επιτροπή στην προηγούμενη θητεία και είμαστε βέβαιοι ότι η έκθεση του συναδέλφου Τάκουλα που όπως είδατε επικεντρώνεται σε τρία πολύ ε, εύστοχα ζητήματα και είναι και ζητήματα επί των οποίων ε, πρέπει να επεξεργαστούμε, θα αποτελέσει τη συνέχεια. Ε, θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες δράσεις που ε, μας αφορούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με την όθηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας ενθαρρύνουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσετε. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική ε, η έκκληση για τη στρατηγική στιγμή στην οποία θα μπορούσαμε να παρέμβουμε για το επόμενο ευρωπαϊκό ε, πρόγραμμα 2017-2020. Να δώσω αμέσως το λόγο στους συναδέλφους που είναι και σκιώδεις συγητές για την έκθεση αυτή. Ο κύριος Νέκοφ ε, που είναι ο πρώτος που ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε και ο Στάβουλα και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι Πιστεύω πως πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν οι πρόσβασης πρόσβαση στο Erasmus Plus. Και ο συνάδελφος μας ανέφερε τη χρηστή ε, διακυβέρνηση, τα κίνητρα και τις ε, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές κτλ. Ε, θα μιλήσω εκ μέρου της κυρίας Μάρλεν Μίτση και ηγήτρια των Σοσιαλδημοκρατών. Ε, η κυρία Μίτση πιστεύει ότι η έκθεση αυτή θα διαδραματίσει σημαντικό ε, ρόλο. Ο αθλητισμός ε, είναι κάτι που ωφελεί πολλού στον κόσμο και αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου είναι και μετά οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ρίο είναι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις οι οποίες μας δίνουν μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τα ωφέλη του αθλητισμού. Και χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό, έτσι ώστε να εμπνεύσουν και ε, μεγάλους και παιδιά να συμμετέχουν σε περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες. Η συμμετοχή των πολιτών στον αθλητισμό επίσης προωθεί την κοινωνική διάδραση και την καλή υγεία. Η προώθηση λοιπόν και η στήριξη του αθλητισμού είναι σημαντική όχι μόνο για την ε, φυσική κατάσταση, αλλά και για τη δυνατότητα που παρέχει να ε, προωθεί το δίκαιο ανταγωνισμό, την αλληλεγγύη, την ε, ανοχή και άλλες κοινωνικές αξίες. Δυστυχώς όταν υπάρχουν μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις βλέπουμε και την άσχημη πλευρά του αθλητισμού, το πώς ε, ε, δηλαδή ένα και περισσότερες φορές ακούμε για περιπτώσεις απάτης, ντόπινγκ, διαφθοράς σε μεγάλες αθλητικές ε, διοργανώσει μεγάλες αθλητικές ε, ομάδες για περιστατικά με τους οπαδούς, ε, με την ασφάλεια και θέματα υγείας, όπως για παράδειγμα η μετάδοση του ιού Ζήκα, αλλά και τρομοκρατικές απειλές. Χρειάζεται λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό, έτσι ώστε οι αθλητικές διοργανώσεις, οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις να είναι ένα υπόδειγμα διαφάνειας χρηστής διακυβέρνησης και ακεραιότητας και να υπάρχει επίσης λογοδοσία και αεφορία. Ελπίζω λοιπόν η έκθεση αυτή να συμπεριλάβει τις προτάσεις καταπολέμησης του ντόπιν ε, και των ε, ουσιών που αυξάνουν τεχνητά τις επιδόσεις των αθλητών. Χρειάζονται ελάχιστα κοινά πρότυπα για τα στάδια, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε οι αγώνες να είναι ε, όσο το δυνατόν ασφαλέστεροι για τους ε, θεατές και επίσης ε, να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός να δοθεί περισσότερη προστασία στους ανηλίκους έτσι ώστε ο αθλητισμός να είναι μια γιορτή. Χρειάζεται επίσης να ολοκληρώσετε, λέει η πρόεδρος, παρακαλώ. να θέλω μισό λεπτό ακόμα. Χρειάζεται λοιπόν δράση έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η διαφθορά και να προωθηθεί η ηθική. Χρειάζεται οικονομική, ε, οικονομικός έλεγχος έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια, ο ίσος ανταγωνισμός και ε, να ε, υπάρχει πρόληψη των παράνομων στοιχημάτων και των στημένων παιχνιδιών. Ο αθλητισμός επίσης ε, έχει οικονομικά ωφέλη και πρέπει να κοιτάξουμε και τι γίνεται με τα δικαιώματα μετάδοσης αθλητικών ε, διοργανώσεων. Διότι μόνο έτσι θα αυξηθεί το ενδιαφέρον και η προθυμία των Ευρωπαίων πολιτών για να φιλοξενήσουν στις χώρες τους αθλητικές διοργανώσεις. Διακόπτει η Πρόεδρος. Και χρειάζεται λοιπόν να, ε, δώσουμε, να στηρίξουμε τα αθλητικά πρότυπα της Ευρώπης. Συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος, πρέπει να σας διακόψω. Ναι, μα έπρεπε να διαβάσω όλη τη δήλωση της ε, συναδέλφου. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή που δείξατε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, να σας υπενθυμίσω ότι θα είστε και υποψήφιος για να είστε μόνιμος εισηγητής για το πρόγραμμα Erasmus+. Έχετε λοιπόν ιδιαίτερε ευαισθησίε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα καταρχάς να πω πως χαίρομαι πάρα πολύ ο, με το ότι ο κύριος Τάκουλα ανέλαβε αυτήν την τόσο σημαντική έκθεση. Ο αθλητισμός είναι πολύμορφος. Είναι η έκφραση της ειρήνης και της ανοχής. Είναι μια αξία ανθρώπινη και για πολλούς ο αθλητισμός είναι τρόπο ζωής. Είναι κάτι θετικό, κάτι καλό. Όμως έχει και ένα άλλο πρόσωπο ο αθλητισμός στην εμπορική του διάσταση. Η οποία εμπορική διάσταση έχει οδηγήσει στη δημιουργία ολόκληρης βιομηχανίας πίσω από τον αθλητισμό. Υπάρχει ολόκληρη λοιπόν οικονομία στην οποία στηρίζονται πολλές θέσεις εργασίας. Ο αθλητισμός επίσης αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του ΑΕΠ. Υπάρχουν πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες ε, καταγράφουν μεγάλα κέρδη από τον αθλητισμό. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω με τους εμπειρογνώμονες και να τους ευχαριστήσω για το ότι ήρθαν εδώ και μας παρουσίασαν τις απόψεις τους. Δυστυχώς ο αθλητισμός έχει και τη σκοτεινή του πλευρά. Τα παράνομα στοιχήματα, τα στιμένα παιχνίδια, διαφθορά και πάνω απ' όλα το ντόπινγκ. Το ντόπινγκ είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε εδώ και πολλά χρόνια να το πολεμήσουμε με διάφορους τρόπους. Το 2008 υπήρχε, ε, δημιουργήθηκε ο διεθνής οργανισμός κατά του ντόπινγκ. Ήμουν μέλος για πολλά χρόνια και προσπαθήσαμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Χρειάζεται όμως να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες και αυτό θα γίνει για παράδειγμα με το να υπάρχουν περισσότερα εργαστήρια που θα διεξάγουν ελέγχους. Στην Ευρώπη υπάρχουν αρκετά από αυτά. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά ε, παραθυράκια στη Ρωσία, για παράδειγμα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα ε, σε πολλούς να ξεφεύγουν από την, ε, τις πολιτικές καταπολέμησης του ντόπινγκ. Πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την ε, καταπολέμηση του ντόπινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η συνάδελφος Νταμάτο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε κυρία Πρόεδρε. Είμαι βέβαιη ε, ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις πολιτικές αθλητισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να προωθήσουμε υψηλότερα επίπεδα προστασίας ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων τις ψυχοσωματικές ε, αξίες που συνδέονται με τον αθλητισμό και γενικότερα την πρακτική του αθλητισμού ως ε, σημείο που ενώνει ε, με πολίτες οι οποίοι έχουν παρελθόν και ιστορία τελείως διαφορετική. Ο αθλητισμός καταρχάς θα πρέπει να ορίζεται και να αναφερόμαστε σε αθλητική παιδεία και να ξεκινά από το δημοτικό σχολείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευσης ε, ε, διδάσκοντες ε, για τον αθλητισμό. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλες δεξιότητες θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση της πολιτείας και θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικών από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά όχι μόνον φαίνεται με το πέρασμα του χρόνου ότι αλλάζουν οι πρακτικές του αθλητισμού και ε, ορισμένες φορές ε, προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να πάμε στη σωστή κατεύθυνση. Ε, στήσιμο παιχνιδιών και κάποιες άλλες κερδοσκοπικές πρακτικές επηρέασαν αρκετά κράτη-μέλη και έτσι έχει χαθεί το «εφαγωνίζεστε» και η αγάπη για τον αθλητισμό πολλών παθιασμένων φιλάθλων πολλές φορές ε, σχετίζονται ε, με τη δράση οργανωμένου εγκλήματος ε, και μαφίας και ορισμένες φορές έχουν διεισδύσει στο σύστημα μόνιμα με τεράστια κέρδη και μέσω παρανόμων στοιχημάτων ή μέσω αντίστοιχης δραστηριότητας. Χρησιμοποιούν ένα χρηματοδοτικό σύστημα σχεδόν εκτός ελέγχου και καταφέρνουν να ε, κάνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες ξεπλήματος, ε, νομιμοποίησης παρανόμων εισόδων και υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί αθλητισμού δηλώνουν ότι αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις ορισμένες φορές απειλούν και εκβιάζουν τους αθλητές ε, και θεωρούν ότι προέχουν ενός πλαισίου. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να προστατεύει ούτως ή άλλως τους αθλητές και να συλλαμβάνει τους δράστες. Ε, ακόμα σήμερα βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κυρώσει την σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χειραγώγηση των αθλητικών εκδηλώσεων. Αντιστοίχω, δεν προβλέπεται ένα σαφέ πλαίσιο δράση που περιλαμβάνει μέτρα τα οποία θα αυξάνουν τη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση των επαγγελματικών αθλητικών συλλόγων και ε, θα έπρεπε να υπάρχει ένα ανώτατο όριο στις αμοιβέ των ε, προπονητών και να υπάρχουν και πειθαρχικές και δεντολογικές επιτροπές ε, των αθλητικών ομίλων. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ανανέωση του αθλητισμού και να υπάρχουν αρχέ οι οποίε θα βρίσκονται στο επίκεντρο τη αθλητική δραστηριότητα. Μόνο αν έχουμε το σθένο να παραδεχτούμε ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε μέχρι τώρα είχαν και κενά και ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τον αθλητισμό και να τον βελτιώσουμε σε όλα τα επίπεδα, θα μπορέσουμε να έχουμε μια ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης. Ένα νέο αθλητικό ε, τρόπο, μια νέα νοοτροπία που θα μας επιτρέπει να δούμε πιο αποτελεσματικά ότι δεν χρειάζεται το ντόπινγκ και στόχο έχει απλώς να μολύνει τη ζωή των αθλητών και τις ε, αξίες που θα έπρεπε να διέπουν την αθλητική δραστηριότητα. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα τα οποία θα ε, παρουσιάσουμε στον εισηγητή και θα συνεισφέρουμε με απτό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο λόγος του συνάδελφο Βέντα, που είναι ε, πρωταθλητής ε, ε, στην Πολωνία, αλλά έπαιξε και στην Πολωνία και στη Γερμανία και στην Ισπανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλες και όλους για τις παρουσιάσεις τους. Ευχαριστώ λοιπόν και ε, βρίσκω πολύ σημαντικά ε, και σχέδιο τον κύριο Τάκουλα που εργάζεται υπέρ της πρόθεση του αθλητισμού. Βεβαίω, ο αθλητισμό μπορεί να συμβάλλει στην ελκυστικότερη παρουσίαση των ευρωπαϊκών αξιών. Ο αθλητισμός μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και στην επίτευξη στόχων εσωτερικής πολιτικής. και στην αναπτυξιακή πολιτική μπορεί πάλι ο αθλητισμός να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Μαζί με τον Επίτροπο Ναύρατσιτς έχουμε εγκύψει στο θέμα αθλητισμός για την ενσωμάτωση ή για την ένταξη στις ε, ε υποδοχής των προσφύγων. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον αθλητισμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αθλητισμό και στις διπλωματικές μας προσπάθειες. Να πούμε ότι ο αθλητισμός παίζει σημαντικό ρόλο και για την προετοιμασία του ανθρώπου, για την περαιτέρω επαγγελματική του ζωή. Μιλήσαμε και ακούσαμε πολλά για την αυτονομία των μεγάλων αθλητικών οργανώσεων. Έχουμε μια οργάνωση τώρα η οποία ασχολείται με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Διεξάγεται αυτό το πρωτάθλημα τώρα και βλέπουμε να λείπει η διαφάνεια. Ελλείψεις βλέπω να υπάρχουν και στην ανάληψη ευθυνών κύριος Τζαμπάσκη και μετά ο επόμενος συναδέλφος. Παρακαλώ να ολοκληρώσουμε γιατί θα έχουμε και την παρουσίαση της μελέτης. Με χαρά παρουσιάζω την γνωμοδότηση εκ μέρους της συναδέλφου μου Μακλάρκιν. Βεβαίως δεν διαθέτω την εγωιτευτική φωνή της ούτε και το εγωιτευτικό παρουσιαστικό της. Ελπίζω ωστόσο ότι θα αρκιστείτε στο άτομό μου. Ο αθλητισμός και ιδίως ο αθλητισμός βάσης είναι σημαντικό θέμα για την συναδελφό μου και χαίρομαι που προωθείτε. Η αρχική πρωτοβουλία που ανέλαβε η ομάδα ECR για την ενσωμάτωση του αθλητισμού σε αυτές τις βασικές πρωτοβουλίες βρίσκω ότι είναι σημαντική. Θέλω λοιπόν να προωθηθούν ορισμένα πράγματα. Στην Έκθεση φύσα του 2011. Αυτή είχε στοχεύσει ιδιαίτερα στον επαγγελματικό αθλητισμό, και ιδίω στο ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω μια έκθεση που να είναι πολύ αθλητική, α το πω έτσι. Δηλαδή να ασχολείται με πολλά αθλήματα. Και αυτό θα πρέπει να είναι ο βασικό στόχο μα. Η πρόταση τη ομάδα ECR θέλει να χρησιμοποιήσει και το πρόγραμμα Erasmus Plus ώστε να διοχετευτούν χρηματοδοτήσει στα αθλήματα εκείνα τα οποία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά προσφέρουν κιόλα και ε, πρότυπο για τους νέου για να μπουν στα αθλήματα αυτά οι νέοι και οι νέε και να παραμείνουν αθλητικά ενεργοί. Αυτά είναι οι απόψεις τη κ. Μακλάρκιν. Ευχαριστώ, λέει η κ. Σόντροβα. Πολλά είπαν οι συναδελφοί μου από τα όσα θα ήθελα να πω και εγώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ενθαρρύνω να προχωρήσει στις δραστηριότητε. της. Οι υποδομές επίση είναι πολύ σημαντικέ. Αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητε υποδομές, πώς να αθληθεί κανείς. Θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνω στο πρόγραμμα να ληφθούν υπόψη και οι αθλητικές υποδομές που πρέπει να δημιουργηθούν και να προωθηθούν. Πρέπει ωστόσο να αντισταθούμε κατά του ντόπινγκ καθώς και κατά του, max, του match fixing συγγνώμη. προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν και να γίνει προσπάθεια και στο ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμα μάλιστα περισσότερο στο παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω εκεί μπορούμε να παίξουμε ένα θετικό ρόλο. Σας ευχαριστώ όλες και όλους και σας ενθαρρύνω, σας αποτείνω λόγια ενθάρρυνσης όλοι εμείς εδώ που ε, είμαστε υπέρ του αθλητισμού είμαστε στο πλευρό σας. Η Πρόεδρος, μήπως έχετε να προσθέσετε κάτι, διότι βεβαίως δεν έθεσαν όλοι οι συνάδελφοι με ερωτήματα, αλλά αν έχετε κάτι που θέλετε να παρατηρήσετε ακόμη, να σας δώσω, δεν έχουμε πολλά λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν έχετε κάτι όμως, ευχαρίστω να σας δώσω το λόγο. Εσείς αποφασίζετε. Αλλά σύντομα. Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα, με συγχωρείτε, διακόπτη η πρόεδρος. Τάκουλα, εσείς θέλετε να μιλήσετε τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα δούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Donc, merci, Madame la Présidente. Donc, j'étais sur le point de dire que je... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να πω ότι δεν θα ε, χρησιμοποιήσω καν το χρόνο μιλίας, αλλά ο κύριος Στάκουλα είπε, εδώ, είπε ότι είναι εδώ για να ακούσει, εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και αυτό θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Ε, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και εγώ εντάξει δεν έχω κάτι να σας πω. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σήμερα αυτή η πρώτη συνέντευξη, συνάντηση κατέδειξε ότι χρειαζόμαστε μια στεναρή πρωτοβουλία, ανοιχτή, και επικεντρωμένη σε κάποιες πτυχές, οι οποίες όμως αποδεικνύεται ότι είναι ουσιαστικές πτυχές για την αξιοπιστία του αθλητισμού και για το μέλλον του. Πολλά από αυτά τα οποία μας είπατε θα είναι πολύτιμα στοιχεία για τον εισηγητή και για τους σκιώδεις εισηγητές και βασιζόμαστε και στην ε, αγαστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ενεργό συμμετοχή σας, αλλά δεν θα πρέπει να ε, ξεχνάμε και τους εμπειρογνώμονές μας κατά την εκπόνηση της έκθεσης, γιατί θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντικός ο διάλογος για μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την παρουσία σας ε, και όλους τους ε, συναδέλφους που ήταν παρόντες, οι οποίοι με ε, βέβαιοι ότι θα παθιαστούν με το θέμα αυτό. Εμένα δεν μου αρέσει ο όρος αθλητισμός ε, και μικρότερα αθλήματα. Θεωρώ ότι όλα τα αθλήματα είναι εξίσου σημαντικά και έτσι θα έπρεπε να αναφέρονται και στην έκθεση. Δεν ξέρω αν είναι εδώ οι ερευνήτριε ήδη στην αίθουσα. Εδώ είναι. Ε, έτσι κατάλαβα καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, την οποία ζητήσαμε, διότι προέκυψε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της διπλής σταδιοδρομίας στον αθλητισμό. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους που είναι ακόμα εδώ να παραμείνουν άλλη μισή ωρίτσα, γιατί αξίζει τον κόπο να ακούσουμε και να συμμετέχουμε σε αυτή την παρουσίαση. Πρέπει να είστε και εσείς εδώ, καθίστε παρακαλώ.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 Eh, λοιπόν, να σας παρουσιάσω αμέσως τις καλεσμένες μας. Έχουμε την ε, καθηγήτρια Λάουρα Καπράνικα ε, και την ε, κυρία Φλάβια Γκουιντότη. Δέκα λεπτά για να ακούσουμε την παρουσίαση και από εκεί και πέρα θα γίνει συζήτηση. Νομίζω ότι μπορείτε να επιλέξετε σε ποια γλώσσα θέλετε να κάνετε την παρουσίαση. Η διαφάνεια ούτως ή άλλως είναι στα αγγλικά. Κάντε όπως νομίζετε κυρία Καπράνικα. Δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο, σας δώσω το λίγο. Λοιπόν, για να είμαι πιο συνοπτική θα τα πω στα Ιταλικά. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε σήμερα να συζητήσουμε το θέμα της ε, εκπαίδευσης και του αθλητισμού και θα το συζητήσουμε από κοινού παρά το γεγονό ότι στην Ευρώπη η εκπαίδευση και ο αθλητισμός ε, είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετοι τομείς, ε, μιλούν τελείως διαφορετική γλώσσα, Ξεχωριστέ γλώσσες και ορισμένες φορές δεν υπάρχουν σημεία επαφής μεταξύ των δύο τομέων. Αναφερόμαστε σε διπλή σταδιοδρομία, διότι Καταρχά εννοούμε την ικανότητα του ατόμου να συνδυάσει μία ή περισσότερε σταδιοδρομίε, στην περίπτωση του αθλητή την αθλητική σταδιοδρομία ή την, και την εκπαιδευτική ή την εργασιακή σταδιοδρομία, διότι δεν επιτρέπουν όλα τα αθλήματα στους αθλητές ε, να συντηρηθούν ε, με τα έσοδα από την αθλητική τους δραστηριότητα. Η παρουσίαση ε, διαρθρώνεται σε 7 σημεία. Οι διαφάνειες είναι αρκετά πυκνέ. Εγώ θα προσπαθήσω να συνοψίσω όσο το δυνατόν περισσότερο αυτές τις πληροφορίες. Δεν θα σταθώ πολύ στο ρόλο του αθλητισμού, τον οποίο ούτως ή άλλως ε, ε, γνωρίζετε όλοι σαφέστατα. Να σας υπενθυμίσω απλώς ότι ανεξάρτητα από την ε, βασική αθλητική εκδήλωση που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες ε, στην Ευρώπη, θα αναφερθούμε και σε πολλά αθλήματα τα οποία δεν ε, προωθούνται και δεν προβάλλονται τόσο πολύ στις, στην καθημερινότητά μας, αλλά απαιτούν μεγάλη αφοσίωση από πλευράς του αθλητή και πραγματικά πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να ε, φτάσει κάποιος και στα υψηλότερα επίπεδα. Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο θα έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε και αυτά τα αθλήματα. Να σας πω ότι ε, Υπάρχει και το πρόσφατο ε, αθλητικό γεγονός των Ολυμπιακών Αγώνων για τους νέους. Αυτό από τη μια δημιουργεί κάποιο ενθουσιασμό αλλά και κάποια ανησυχία όσον αφορά την προστασία και την ανάπτυξη του νέου αθλητή. Ο αθλητής ε, αναγνωρίζεται ε, πάντα είναι πολύ σημαντικό αυτό και μέσω της εθνικής του αναγνώρισης αλλά και για τις κοινωνικές πτυχές αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί αθλητές ε, διαδραματίζουν και πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, κοινωνική ζωή στη συνέχεια ως πολιτικοί ή ως προπονητές. Ε, αθλητές οι οποίοι κατάφεραν να συνδυάσουν την ε, εκπαίδευσή τους, την καταρτισή τους με ε, και την εκμάθηση των δεξιοτήτων για τη ζωή αργότερα ε, μπορούν στη συνέχεια να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Μια άλλη πτυχή είναι το γεγονός ότι οι δεξιότητες ε, που προκύπτουν από τον αθλητισμό σε γενικές γραμμές είναι κληρονομιά των κρατών μελών, που σημαίνει ότι εμείς έχουμε μία σειρά από ε, και ο όρος αθλητισμός και εκπαίδευση χρησιμοποιούνται μεν ε, ο ένας στη θέση του άλλου, αλλά υπάρχουν κάποιες ουσιαστικές διαφορές. Κάποιες χώρες έχουν ε, μια μορφή αθλητισμού ε, και πρόσβαση στον αθλητισμό που διευκολύνεται από το σχολείο ήδη, ενώ σε άλλες χώρες ε, στο δημοτικό σχολείο δεν υπάρχει μάθημα φυσικής αγωγής. Επομένως ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε. θεωρώ ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε ίσως να υπάρχει δυνατά να ε, εκμεταλλευτούμε τη μεγάλη αυτή ευκαιρία της ποικιλομορφία και να βρούμε νέες και καινοτόμες ε, λύσεις ε, και από πλευράς αθλητισμού και παιδείας ώστε να προσπαθήσουμε να μεγενθύνουμε και να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή κουλτούρα του αθλητισμού. Αυτή τη στιγμή το φαινόμενο αθλητισμός δεν είναι σαφές, γιατί επειδή δεν είναι σαφής οι όροι δεν είναι σαφείς ούτε και οι δεξιότητες και οι ευθύνες και επομένως δεν έχουμε ε, στατιστικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να ορίσουμε το φαινόμενο στο σύνολό του. Μία άλλη πτυχή την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το γεγονός ότι το άτομο, είτε είναι αθλητές είτε όχι, είναι ένα ενιαίο σύνολο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όσο τον αναγνωρίζουμε ως αθλητή είναι σαν να ξεχνάμε ότι έχει παρελθόν γιατί ο αθλητής δεν δημιουργείται ξαφνικά αλλά το, το χτίζεις. Ε, ο πρωταθλητής ε, για να τον κατανοήσουμε θα πρέπει να κατανοήσουμε όλα τα στάδια από την πρώτη του εισαγωγή στον αθλητισμό στην ανάπτυξή του, στην ε, στήριξη του ταλέντου του μέχρι την αθλητική σταδιοδρομία η οποία θα μπορούσε να διακοπεί ανα πάσα στιγμή και λόγω τραυματισμών. Ε, πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε στο σύνολό του. Θα πρέπει ε, λοιπόν να το εξετάσουμε αυτό και να κατανοήσουμε έτσι τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει ε, εάν σε έναν αθλητή στον οποίο έχουμε στερήσει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί ως πολίτης και να εκπαιδευτεί και ως άτομο τι πρέπει να κάνουμε για να το ξαναεντάξουμε στο κοινωνικό πλαίσιο. Αυτή είναι μια εξαιρετική διαφάνεια που ε, ε, έφτιαξε η Ομάδα Ανθρωπίνων Πόρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά την κατάρτιση. Όταν οι ανάγκες του αθλητισμού και της παιδείας αυξάνονται περνώντας από το δημοτικό σχολείο στο γυμνάσιο και στη συνέχεια ε, στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο, ο αθλητής ε, μπορεί να επιλέξει και ή επιλέγει να συνεχίσει και να ακολουθήσει το ταλέντο του και ορισμένες πολύ συχνά να θυσιάσει την εκπαίδευσή του και αυτή είναι συχνά μια επιλογή των ανδρών ή επιλέγει να εκπαιδευτεί για το μέλλον επομένως εγκαταλείπει το αθλητικό του ταλέντο προ όφελο ε, τη εκπαίδευσή του. Και αυτή είναι μια επιλογή που κάνουν κυρίω οι γυναίκε, που σημαίνει ότι εμεί στον αθλητισμό χάνουμε πάρα πολλού πόρου ε, από πλευρά γυναικών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι φρικτό και αν δεν το υποστηρίξουμε και σε επίπεδο διακυβέρνηση, ε, και δυστυχώ η διακυβέρνηση, λυπάμαι που θα στο λέω, είναι υπέρ του ανδρός, δύσκολα μπορούμε να αντιληφθούμε το φαινόμενο. Υπάρχουν διάφορα ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν σε αυτή τη διπλή σταδιοδρομία του αθλητή. Ο αθλητής είναι το κεντρικό πρόσωπο, ε, τα κίνητρά του είναι κεντρική σημασία, αλλά υπάρχουν και όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το μικρό κόσμο του αθλητή. Υπάρχουν οι γονείς, οι προπονητές, ε, οι διευθυντές, οι συνάδελφοι, οι συμμαθητές στο σχολείο, οι συναθλητές. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και εδώ έχουμε και την οργανωτική διάσταση. Το σχολείο όπως είναι οργανωμένο και ε, ο αθλητισμός και όταν δεν υπάρχει συνομιλία ο αθλητής ε, βρίσκεται ε, ουσιαστικά στο μέσο και αυτό δεν είναι σωστό. Ε, και μετά υπάρχουν εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Εσείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε, είστε αυτοί οι οποίοι μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη χιονοστιβάδα και να προσπαθήσετε να επηρεάσετε και να συστήσετε θα μπορούσαμε να πούμε διότι προφανώς οι πολιτικές είναι από εκεί και πέρα αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα άτομο, αλλά για ομαδική δουλειά. Εγώ ε, προέρχομαι από τα ομαδικά αθλήματα και κατανοώ πώ είναι τα αθλητικά, ομαδικά αθλήματα. Και στο πανεπιστήμιο η έρευνα είναι μια ομαδική δραστηριότητα και η διπλή καριέρα, η διπλή σταδιοδρομία είναι ακόμα περισσότερο ομαδική δραστηριότητα, διότι συνενώνει διάφορου τομεί. Υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα σε κάποιες χώρες, στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στην Γαλλία, στην Ισπανία και στην Αγγλία. Ε, φανταστείτε ότι στην ε, Γαλλία και στην Αγγλία τα περισσότερα αθλητικά μετάλλια τα έπαιρναν, ολυμπιακά μετάλλια τα έπαιρναν αθλητές που είχαν διπλή σταδιοδρομία. Ήταν και φοιτητέ και ε, αθλητές ε, με μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχουν όμως χώρες που δεν έχουν την ίδια προσέγγιση, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος για να επιλύσουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και να ε, τροποποιήσουμε να αλλάξουμε το ε, περιορισμένο όριαμά μας. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε και κατάλληλη δικτύωση. Και εδώ ε, πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι διότι είμαι πρόεδρος της ΕΑΣ που είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο του Αθλητή ως Φοιτητή το οποίο ιδρύθηκε το 2004 ε, Ευρωπαϊκό Έτος Αθλητισμού και κάθε χρόνο διοργανώνει μία ετήσια διάσκεψη στην οποία συναντούνται όσοι ε, διοργανώνουν και υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα προκειμένου να συζητήσουν και τις εμπειρίες τους αλλά και τα αποτελέσματα των διαφορών εμπειριών. Εδώ σε αυτό το δίκτυο έχουμε και αθλητικούς συλλόγους αλλά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και είναι ε, ένας χώρος ε, διαλόγου με τελείως διαφορετική γλώσσα. Φέτο θα γίνει εκδήλωση στο Ροβανιά εμείς, στο σπίτι του Αγίου Βασίλη και από 15 έως 17 ε, Σεπτεμβρίου θα είμαστε εκεί και θα κάνουμε μια λίστα με τις επιθυμίες μας. Οι πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετικές. Ε, το 2010 έγινε μια ταξινόμηση σε μια μελέτη που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και Καθορίσαμε τέσσερις κατηγορίες, χώρες ε, στις οποίες υπάρχει κεντρική ρύθμιση και χώρες στις οποίες δεν υπάρχει καμία διευκόλυνση και ο φοιτητή αθλητή είναι υποχρεωμένος να διαπραγματεύεται μόνο του την ιδιαίτερη κατάστασή του και ορισμένε φορέ να κρύβεται ή να λαμβάνει αποφάσει ε, με απομονωμένο τρόπο, αλλά η κατάσταση αυτή εξελίσσεται συνεχώς, διότι υπάρχουν κάποιες χώρες, όπως η Αυστρία για παράδειγμα, ε, που θεωρούνται ε, μία από τις χώρες που δεν έχουν νομοθεσία από του θέματος και έχουν ήδη προσαρμοστεί. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε αν την τάση αυτή την ακολουθούν και άλλες χώρες. Υπάρχουν διάφορα συστήματα και αν ε, και ε, τα έχουμε κατηγοριοποιήσει σε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες, δεν σημαίνει ότι κάθε χώρα έχει το ίδιο σύστημα. Απλώς λέμε ότι το κράτος ε, με συγκεκριμένη νομοθεσία ρυθμίζει την κατάσταση. Επομένω, η διπλή σταδιοδρομία εξαρτάται και από το εκπαιδευτικό σύστημα τη κάθε χώρα, ε, τι πολιτικέ για τον αθλητισμό τη κάθε χώρα και το συγκεκριμένο άθλημα. Διότι, για παράδειγμα, στα ε, αθλητικά παιχνίδια σε σχέση με, τις, ε, με τα αθλήματα που είναι αθλήματα αγώνων, ή αθλήματα όπως το box ε, έχουν τελείως διαφορετικό ακόμα και τρόπο προπόνησης. Επομένως όλα αυτά έχουν σχέση και με τη διπλή σταδιοδρομία του φοιτητή αθλητή. Μια άλλη πτυχή είναι το γεγονός ότι ο φοιτητή αθλητής που αναγνωρίζεται είναι κάτι τελείως διαφορετικό σε κάθε χώρα ένας φοιτητής, αθλητής θα μπορούσε ίσως να θεωρείται ότι έχει κάποια, δικαίωμα σε κάποιες υπηρεσίες σε μια χώρα και αντίστοιχα ο αντίπολός του στο πρωτάθλημα για παράδειγμα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπορεί να μην τη χάνει της ίδιας αναγνώρισης. Επομένως πρέπει να υπάρχει ένας σαφής ορισμός για το ποιος είναι αυτός ο αθλητής φοιτητής, ε, ποιες είναι οι διάφορες φάσεις ανάπτυξης μέχρι να γίνει ε, αθλητής, φοιτητής ε, που κάνει πρωταθλητισμό και ε, με βάση ποια κριτήρια θα θεωρείτε ότι είναι επιλέξιμος για να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία. Μία άλλη πτυχή είναι το γεγονός ότι ακόμα και η αθλητική και εκπαιδευτική πορεία του κάθε αθλητή φοιτητή διαφέρουν ανάλογα με τον καθένα. Χρειάζεται λοιπόν πολύ μεγάλη ευελιξία και από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολύ συχνά το εκπαιδευτικό ίδρυμα συχνά έχει μόνο σήμαντη κατεύθυνση και πολύ δύσκολα μπορούμε να βρούμε εναλλακτικέ λύσει, αλλά και ε, ο αθλητικός οργανισμός αντίστοιχα. Και υπάρχει και μια άλλη πτυχή που θα έπρεπε μάλλον να υπάρχει, υπάρχει μια διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της εξέλιξης του φαινομένου. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαδικασία, δεν υπάρχουν ορισμοί, δεν υπάρχουν μέσα, δεν υπάρχουν κατάλληλα όργανα, διότι μεταξύ άλλων τα όργανα πρέπει να είναι εξωτερικά, διότι αν είναι εσωτερικά, εντός του εκπαιδευτικού συστήματος ή του αθλητικού συστήματος, ε, μπορεί ταυτόχρονα να αποτελούν και αντικείμενο χειραγώγησης. Ε, η άλλη ουσιαστική πτυχή είναι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο δίνονται πιστοποίησεις. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες έχουν υλοποιηθεί 18 έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια είναι ακόμα εν εξελίξη. Ε, κανένα από αυτά δεν αφορά την παρακολούθηση. Η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται με πιλωτικά προγράμματα, διότι είναι τελείω διαφορετικέ οι διάφορες καταστάσεις. Και φυσικά ελπίζω να το συμπεριλάβετε και αυτό στο θεματολόγιο σας κάποιες άλλες πτυχές, διότι βλέπω ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Είναι κάποιες νέες μελέτες οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει και μία μελέτη για τις ελάχιστες απαιτήσει ε, για αυτή τη διπλή διοδρομία και τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται και αυτό που έχει σημασία είναι ότι και πάλι αναφέρεται ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε στην κατάλληλη παρακολούθηση. Σας επισημαίνω λοιπόν αυτή την πτυχή κάτι τελευταίο. Ο αθλητής μετανάστης που είναι αυτός ο οποίος ε, πρέπει να φύγει για ένα διάστημα, είτε για προπόνηση, είτε για αθλητικές εκδηλώσεις ε, και είναι ένα πολύ συγκεκριμένος ε, αθλητής, ε, τον οποίο ε, πολύ συχνά τον χάνουμε, διότι υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση από το Αμερικανικό σύστημα που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ένταξης αθλητών φοιτητών. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε και εμείς να διευκολύνουμε τους δικούς μας τους φοιτητέ και εδώ δεν θα μακρηγορήσω, τα είπατε κι εσεί το Erasmus Plus για τον αθλητισμό, αυτό θα έπρεπε να κάνει και θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ε, προγράμματα ε, εξειδίκευσης τα οποία θα δίνονται απλώς και μόνο σε εθνικούς φοιτητές. Εάν κερδίσει ένα εθνικό μετάλλιο ένα δανό φοιτητή σε σχέση με έναν Ιταλό, φυσικά μπορεί να υπάρχει πρόβλημα εθνικισμού, αλλά στην Ευρώπη είμαστε. Επομένω θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη και σε αυτή την πτυχή και να πείσουμε και τα κράτη-μέλη προσφέροντα κίνητρα, προσφέροντα ε, ε, κάποιες ε, ε, σκέψεις και συμβουλές. Ε, δεν ξέρω τι ακριβώ θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα μπορούσαμε να το επεξεργαστούμε. Τελευταία πτυχή είναι οι αθλητικές δεξιότητε. Εδώ και πάλι έχουμε μεγάλη ποικιλία. Ο πανεπιστημιακός κλάδος εντάχθηκε πρόσφατα και πολύ συχνά οι ομοσπονδίες δεν αναγνωρίζουν τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια δεν αναγνωρίζουν τις ομοσπονδίες. Σας μιλώ ως καθηγήτρια ε, σε ένα ε, τμήμα ε, αθλητή αθλητικών δικαστών για τον αθλητισμό. Ε, δεν είμαστε εχθροί, θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για να βελτιωθοποιήσουμε το σύστημα και το σύστημα θα πρέπει να έχει ένα, ένα ελάχιστο κοινό παρελωμαστή ε, με έναν άλλο τρόπο. Και μια ακόμα πτυχή, και εδώ και πάλι χρειαζόμαστε παρακολούθηση. Δεν έχουμε στοιχεία. Η Βουλγαρία και η Ιταλία, ε, η Ιταλία για παράδειγμα έχει έναν τρίτο οργανισμό, την Alma Laura, η οποία παρέχει ε, πληροφορίες όχι μόνο για τους πτυχιούχους, αλλά και για τη σταδιοδρομία τους στη συνέχεια και υπάρχει και η Πορτογαλία και η Σλοβενία που έχουν τελείως διαφορετικά συστήματα η μία από την άλλη αλλά πολύ καλά. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι προβλέπει μία σειρά ε, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση που πρέπει να αναγνωριστεί και σε σχολικό και πανεπιστημιακό επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο θα πρέπει να επεξεργαστείτε και δυστυχώς ακόμα δεν άκουσα τίποτα από αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε ποια είναι τα σαφή όρια μεν, αλλά η αναγνώριση της ε, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ρωτήστε πρώην ε, αθλητέ, πρωταθλητέ που έχουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Είναι μία από αυτές τις πτυχές λοιπόν που ελπίζω ότι θα μπορέσετε και θα θελήσετε να επισημάνετε. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να βρούμε κοινού ορισμούς. Δεν υπάρχει σωστός ορισμός, πρέπει να συμφωνήσουμε λοιπόν επί των ορισμών ή τουλάχιστον επί των βασικών ορισμών. Από εκεί και πέρα ο καθένα μπορεί να χτίσει οτιδήποτε με βάση αυτούς. να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες απαιτήσει, να υπάρχει ε, δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τα πράγματα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια εναρμόνιση στοιχείων και εδώ και πάλι ελπίζω ότι θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια πιλωτικά προγράμματα για κάθε τύπο αθλήματος εγώ προτείνω κάποια με την ε, Συνομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, για παράδειγμα, ώστε να ξεκινήσει, να ανοίξει ένας δρόμος, όχι να έχουμε μια λύση πανάκια για τα πάντα και να υποστηρίξουμε τα εθνικά δίκτυα και διεθνή δίκτυα. Να υποστηρίξουμε και τις διεθνείς συμφωνίες και να υπάρξουν ε, ειδικά προγράμματα αφιερωμένα στους ε, φοιτητές αθλητές. Και επίσης να υπάρχουν και επιστοποιητικά ποιότητας για ε, συλλόγους, ομοσπονδίες, πανεπιστήμια και οποιοδήποτε άλλο. Θα πρέπει να υπάρχει μια προνομιακή σχέση που θα μπορούσε να είναι σημαντική. Και με αυτό είμαι στη διάθεσή σας, εγώ και η κυρία Γουιντότη ό,τι και να θέλετε να ρωτήσετε είμαι στη διάθεσή σας ή από εκεί και πέρα στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας, κυρία Καπράνικα. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία αποδεικνύουν ότι πράγματι πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο πλαίσιο. Αυτό μας το προσφέρει η έρευνά σας με σαφή τρόπο και η εμπειρία σας, ε, πολλαπλή εμπειρία σας, σε ποιο άθλημα ήσασταν? Στο μπάσκετ, ναι, το κατάλαβα. Ε, ήσασταν σε ομάδα. Και εγώ ήμουνα ε, σε μια ε, εθνική γυναικών. Εγώ όχι, λέει η κυρία Καπράνικα, έκανα άλλη επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι τα ομαδικά αθλήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, ιδίω για τι γυναίκε. Εσείς λοιπόν με αυτή την πολλαπλή σας ιδιότητα έχετε και την πανεπιστημιακή ιδιότητα, την αθλητική ιδιότητα και με το δίκτυο αυτό στο οποίο συμμετείχετε μας είπατε λίγες ελλείψεις που υπάρχουν και νομίζω ότι μέσω αυτής της έκθεσης τάκουλα η πτυχή αυτή θα μπορούσε να συμπεριληφθεί διότι ε, πρόκειται για ε, πολύ σημαντικά στοιχεία ε, αφορούν και την προσβασιμότητα αλλά και την ακαιρεότητα και την κατάλληλη διαχείριση. Είναι λοιπόν εγκάρσια τα θέματα θέματα αυτά. Δεν είναι εδώ βέβαια ο κύριο αλλά θα του το διαβιβάσουμε. Οι συνάδελφοι θέλουν το λόγο για αυτή τη μελέτη, έχουν κάποιε ερωτήσει. Ε, κυρία Εγώ έχω πτυχίο στις ε, κινητικές επιστήμες. Υπάρχουν κάποιες βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη όσον αφορά την ε, φυσική αγωγή, τις βασικές δηλαδή δεξιότητες στα δημοτικά σχολεία και στους αθλητικούς συλλόγους. Να υπάρχει δηλαδή φυσική αγωγή ε, και ε, από εκεί και πέρα να υπάρχουν και κάποια πτυχία για αυτούς που πηγαίνουν σε αυτά τα βασικά ε, μαθήματα αθλητισμού, ακόμα και ε, κάθε Σαββατοκύριακο. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο? Έχετε κάποια ερώτηση? Σύντομος. Ε. Θα είμαι σύντομος. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Γι' αυτό βρισκόμαστε και εμείς εδώ. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες τις πληροφορίες αυτές, γιατί και Προσωπικά, εγώ ως νέος ε, είχα εμπλακεί και επαγγελματικά. Δηλαδή έπαιξα handball επαγγελματικά, μετά έγινα και προπονητής και στη διάρκεια της αθλητικής μου σταδιοδρομίας πάντοτε προσπαθούσα να αναμειγνύομαι και στο κοινωνικό πεδίο. Αυτό μου έδωσε πολλά σημαντικά διδάγματα για το πώς μπορώ να συμμετάσχω και στις διάφορες τοπικές κοινότητες. Και λοιπόν ε, επαγγελματίας αθλητής και μετά ως προπονητής, αλλά και αργότερα ανέπτυξα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, αλλά και ε, δίδαξα ε, motivation στον αθλητισμό. Άρα πρέπει κανείς να έχει υπόψη ότι οι διπλές σταδιοδρομίες είναι σημαντικές για τους αθλητές, όχι όμως μόνο για την πανεπιστημιακή κατάρτιση, αλλά και για πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε ένα δυναμικό το οποίο μπορούμε μετά να αναπτύξουμε με διαφορετικούς τρόπους. Είναι κρίμα, ίσως τώρα είναι αργά, ενώ είναι προχωρημένη η ώρα, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να μιλήσουμε και για αυτά τα πράγματα και στα πλαίσια του έρασμος συν Ευχαριστώ πολύ πάντως για την παρουσίασή σας και τουλάχιστον εμένα με ικανοποίησε απολύτως. Θα προσπαθήσω να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Σαφώς και είναι πολύ σημαντική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι άρτια καταρτισμένοι. Αυτό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση που ρώτησε η Ιταλίδα Ευρωβουλευτέ. Αντιλαμβάνομαι τι εννοείται. Πρόκειται για ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα που αφορά την Ιταλία. Και εγώ είμαι καρπό αυτού του προβλήματο. Καταλαβαίνω απόλυτα ποιο είναι το πρόβλημα. Πρέπει όμω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχουν εξαιρετικέ πρακτικέ. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, υπάρχει μάθημα φυσική αγωγή για τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο. Υπάρχει ένα σύστημα αλλά δεν είναι απαραίτητα το ίδιο σύστημα αυτό το οποίο θα πρέπει να υιοθετήσουμε. Πρέπει όμως να το μελετήσουμε. Η άλλη πτυχή είναι ότι στην Ιταλία, για παράδειγμα, έγινε ένα πρώτο πρόσφατο έργο με τη Φερέρο, μία συνάδελφός μου, υλοποίηση ένα πρόγραμμα με πτυχιούχους σε κινητικές επιστήμες και τώρα αυτό το πρόγραμμα έχει μεταφραστεί σε τρεις γλώσσες ε, και λέγεται το πρόγραμμα Enjoy Your Moving. Ε, υπάρχουν λοιπόν πολύ ωραία προγράμματα σε πολλές χώρες. Όσον αφορά τώρα την κατάρτιση των ηθινών, των προπονητών, των εκπαιδευτών, ε, όλων αυτών των κατηγοριών ε, ε, που προσπαθήσαμε να μελετήσουμε και με μια μελέτη που έγινε πρόσφατα και που θα δημοσιευθεί εντός ε, ολίγου, ε, δεν υπάρχει καμία συνεκτικότητα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει η ίδια μορφή εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε λοιπόν να κατανοήσουμε ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσει και θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση εάν έχουμε άτομα με παιδεία και από αθλητική σκοπιά αλλά και από ε, πανεπιστημιακή σκοπιά, αλλά όχι μόνο πανεπιστημιακή παιδεία. Ε, μπορεί να είναι και μια σχολή επαγγελματική κατάρτιση. Ε, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αρκεί να είναι καταλήλου επίπεδου. Και αυτό φυσικά πρέπει να προσφέρει και δεξιότητε. Αυτό είναι ο βασικό στόχο κατά την άποψή μου bi se navezal ravno na zadnje vprašanje. Tudi eh, o tem je govoril. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω ε, την ερώτηση του κυρίου Βέντα. Ο κύριος Βέντα μίλησε για τη διπλή σταδιαδρομία και πώς οι αθλητές μπορούν να σπουδάσουν ταυτόχρονα και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε βέλτιστες πρακτικές. Ε, στη Σλοβενία έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα των πρακτικών. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στα σχολεία, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τους αθλητές. Υπάρχουν δηλαδή ε, αθλητικά γυμνάσια, αθλητικά λύκεια. όπου μπορούν οι μαθητές να σπουδάσουν και να ακολουθήσουν αθλητική σταδιοδρομία ταυτόχρονα. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να είναι πάρα πολύ ευέλικτο και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να δίνει τη δυνατότητα αυτής της διπλής σταδιοδρομίας. Ευχαριστώ. Ναι. Σίγουρα το ενδιαφέρον για αυτή την έρευνα είναι πολύ μεγάλο. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι θα έχουμε μία ακόμα ευκαιρία να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, διότι μόλις ε, παρουσιάστηκε το θεματολόγιο για τις δεξιότητες. Και εκεί Σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον από εμά ε, για το θέμα της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων γενικότερα να ε, αναφερθούν και επίσης αυτό που είναι σημαντικό ε, και θα έπρεπε να γνωρίζετε είναι ότι τα λεγόμενα soft skills ε, θα πρέπει να αναγνωρίζονται σήμερα. Είναι λοιπόν άλλη μια ευκαιρία να συμπεριλάβουμε και αυτές τις δεξιότητες οι οποίες ε, προέρχονται και από αυτή την αθλητική εμπειρία θα μπορούσατε ίσως να μας πείτε και την άποψή σας ε, τη δεδομένη ε, στιγμή. Το άλλο θέμα είναι το θέμα της παρακολούθησης. Είπατε ότι έγιναν πολλές συστάσει από αυτού. Ε, θα θέλαμε να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό, με ποιο τρόπο. Διότι υπάρχει και τόσο διαφορετική διαχείριση των αθλητικών εκδηλώσεων του αθλητισμού ε, για να μπορέσουμε να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία θα είναι πολύ περίπλοκο. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι ότι εμείς στη χώρα μας, ίσως και σε άλλες χώρες, έχουμε εμπειρία ε, αθλητών ε, στο στρατό στη συνέχεια. Υπάρχει και εκεί διπλή σταδιοδρομία. Ήλπιζα, για παράδειγμα, να είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Μάλλον κάνω λάθος. Σε άλλε χώρε δεν υπάρχει. Και κάτι τελευταίο, ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το δίκτυο στο οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, το ΕΑΣ. Υπάρχουν έγγραφα του δικτύου που θα μπορούσαν ίσως να κάνουν και κάποιες προτάσεις ε, για να δούμε και τι πλαίσιο θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ε, αυτό το οποίο μας απομένει είναι πολλά διότι νομίζω ότι δεν θα πρέπει να χάνονται οι αθλητές. Αυτό που είπατε για τις γυναίκες είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν θα πρέπει να χάσουμε και τη δυνατότητα να έχουμε αθλητές που αφού σταματήσει η επαγγελματική τους δραστηριότητα ως αθλητές ε, ε, να μην έχουν κάτι να κάνουν. Θα πρέπει ήδη να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ ε, πανεπιστημίων και αθλητισμού μετά από την πιο ισχυρή νομική βάση που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας ε, ε, μπορούμε να ζητήσουμε και μεγαλύτερη αναγνώριση του αθλητισμού. Ο Επίτροπος ε, είναι αρμόδιος και για τον αθλητισμό και για την παιδεία και ο αθλητισμός για πρώτη φορά περιλαμβάνεται και στο Erasmus+. Επίσης να σας πω ότι... Φοιτητέ ε, που ε, αθλούνται κιόλα μπορούν κάλλιστα να συμμετέχουν και στο Εράσμους. Αλλά εδώ αναφερόμαστε στους αθλητές βέβαια. Θα τις έχουμε υπόψη. Δύο πράγματα θα ήθελα να πω. Γνωρίζω ότι η Σλοβενία είναι εξαιρετική η σχέση μου με το Πανεπιστήμιο της Λουμπιάννα και ε, ε, καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε για το Λύκειο. Ε, δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι για το Πανεπιστήμιο και όσον αφορά τα life skills υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βιβλιογραφία και το Joint Moving είναι μεγάλο τμήμα αυτού. Προσπαθούμε τώρα με κάποιε ομοσπονδίε μπάσκετ να δούμε εάν μπορούμε να ελοπίσουμε κάποια πράγματα και παρουσιάσαμε και ένα πρόγραμμα πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, συνεργασία και εταιρική σχέση. Θα δούμε από εκεί και πέρα αν θα γίνει δεχτή η πρότασή μας, ε, γιατί υποβάλαμε μια πρόταση για ένα πρόγραμμα. Στο Κίμη Σλοβένικα έχουμε γράψει και μία μελέτη που εξηγεί τι είναι το ΕΑ στο δίκτυό μας και επίσης να σας πω ότι υπάρχει ε, μία κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται Healthy Diet and Healthy Life Δυστυχώ, βέβαια να σας πω ότι υπάρχουν τρεις πυλώνες. Στον ένα υπήρχε η φυσική δραστηριότητα που ήταν πολύ περιορισμένη όμως. Στο δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα δεν αναφέρεται τίποτα. Εγώ ασχολήθηκα με τον πρώτο πυλώνα. Ε, αναπτύξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο πλαίσιο στο οποίο υπάρχει και το θέμα της διαχείρισης και η διπλή σταδιοδρομία και πολλά άλλα πράγματα. Και Ίσως θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει για την Επιτροπή σας, θα σας στείλω και την επιστημονική μελέτη, αν θέλετε μπορούμε να τη συζητήσουμε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι στο δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα δεν υπάρχει τίποτα γιατί αναφερόμαστε μόνο στη διατροφή, τρόφιμα, διατροφή, δίαιτα κλπ. Πολύ ωραία, εγώ συμφωνώ, ε, πολύ σημαντικό αυτό, αλλά αν αναφερόμαστε σε φυσική δραστηριότητα, σε μια ε, υγιή και δραστήρια ζωή, θα πρέπει να αναφέρεται και ο αθλητισμός. Εδώ αναφερόμαστε στον ε, αθλητισμό και στη φυσική δραστηριότητα και πώς κάποιες φορές είναι το ένα και το αυτό και κάποιες φορές είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο αθλητισμός λοιπόν που θα έπρεπε να είναι μια κοινή γλώσσα, τελικά μιλάει πάρα πολλές γλώσσες και ορισμένες φορές και διαλέκτους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση σα. πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ πολύ και σα ευχαριστούμε και που περιμένατε λίγο γιατί σα καθυστερήσαμε. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσω, αλλά να σας πω ότι η επόμενη συνάντησή μας είναι στις 13 Ιουλίου 9 με 12.30 και 3 με 6.30 και 14 Ιουλίου τελευταία συνεδρίαση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές 9 με 12.30. Η πρόεδρο ευχαριστεί τους Ερμηνείς, ευχαριστούμε και τους συναδέλφου που έμειναν εδώ μέχρι τέλους, ευχαριστώ και τη Γραμματεία και ε, σας ευχαριστώ την προσοχή. Ακόμα και αν είναι Ιούλιο, πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Σα ευχαριστώ πολύ.